chers bonjour. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώ ήρθατε. Ξεκινάμε το πρώτο σημείο στη μερίσια διάταξη, ανταλλαγή απόψεων με τους Ευρωπαίους συντονιστές των διαδρόμων των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Θα μιλήσουμε για, τις, ε, για τους θαλάσσιους αυτοκινητοδρόμους και τη διαχείριση της, ε, των επιβατών στους σιδηροδρόμους. Γεια σας κυρία Γκραπίνη. Είναι δύο οριζόντιες προτεραιότητες όπως ξέρετε, δίπλα από τους ε, διαδρόμους του κεντρικού δικτύου που βρίσκονται στο κέντρο της πολιτικής για τα Τέντη. και υπάρχει επιδότηση αυτών των προγραμμάτων ε, με ουσιαστική συγχρηματοδότηση. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε την πρόοδο που έχει γίνει στους τομείς αυτούς με τους υπεύθυνους συντονιστές. Έχω την χαρά και την τιμή να έχω εδώ τον κύριο Μποντεβίγκ που είναι υπεύθυνο για τις θαλάσσιες οδούς, τους θαλάσσιους αυτοκινητοδρόμους και τον κύριο Ρούτε που είναι υπεύθυνο για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης των, της κυκλοφορίας στους συντηροδρόμους. Καλή χρονιά παρεμπιπτόντος υγεία και χαρά. Σήμερα είσαστε εδώ για να μας εξηγήσετε την κατάσταση. Θα ξεκινήσουμε με εσάς κύριε Μποντβίγκ. Έχετε 7 λεπτά για να μας παρουσιάσετε το που έχουμε φτάσει σε αυτό το θέμα των ε, θαλάσσιων αυτοκινητοδρόμων. Πάνω και από 20 χρόνια ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Κάποια στιγμή πρέπει να επιταχύνουμε, γιατί μια και έχουμε και το πρόβλημα της κλιματικής, της αύξησης θερμοκρασίας ε, του πλανήτη, ίσως είναι μία από τις λύσεις για να λύσουμε το πρόβλημά μας. Ευχαριστώ, αγαπητοί ευρωβουλευτές. Είναι χαρά μου να είμαι εδώ με τη νέα μου ιδιότητα του Ευρωπαίου Συντονιστή για τους θαλάσσιους αυτοκινητοδρόμους, μία από τις οριζόντιες ε, προτεραιότητες του ΤΕΝΤΗ για πέντε χρόνια. Ήμουν ε, Ευρωπα... Ευρωπαίος ε, συντονιστής ε, σε ένα από τους διαδρόμους Βαλτικής Αδιατικής, ένα τεράστιο project και επειδή έχω ασχοληθεί με τους διαδρόμους και με τις οριζόντιες αυτές προτεραιότητες, έχω καταλάβει τις, τα ωφέλη από τις οριζόντιες αυτές προτεραιότητες που θα προκύψουν από την ανάπτυξη των δικτύων αυτών των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Ε, είναι σημεία σύνδεση των συνδυασμένων μεταφορών. Ε, έχουμε τις θαλάσσιες οδούς, ε, όπου εκφορτώνονται και φορτώνονται εκατομμύρια φορτώ, εμπορεύματα και είναι ένα τεράστιο εργαλείο για να βοηθήσουμε την αποσυμφόρηση των, υποδομών των θαλάσσιων αυτοκινητών δρόμων υποστηρίζουν το εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο και την ανταλλαγή προϊόντων μεταξύ ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και τριτών χωρών. Έχει θετική επίπτωση στην προσπελασιμότητα των περιφερειακών ε, περιοχών και αυτό μας βοηθάει γιατί έτσι έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών στην Ευρώπη. Ε, επίσης έχουμε και το Connecting Europe Facility, το SEF, ε, και με αυτόν τον τρόπο συνδυάζουμε λιμάνια, ε, συνδέονται διάφορα λιμάνια από διάφορες χώρες και έτσι ε, επιτυχάνουμε την προσθέμενη αξία. Από την άλλη πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν ήταν εύκολα αυτά τα project, ήταν, είναι περίπλοκο γιατί πρέπει να το συνδυάσουμε με τις ε, χρηματοδοτικές προτεραιότητες του ΣΕΦ. Καταρχά, υπάρχουν περιορισμοί λόγω των κριτηρίων επιλεξιμότητα. Μπορούμε όμως στο μέλλον να βελτιώσουμε την κατάσταση των διαδρόμων αυτών. Χρειαζόμαστε στρατηγικούς στόχους για να υπάρχει καλύτερη διασύνδεση με τους διαδρόμους και να δημιουργήσουμε μια πραγματικά ε, θαλάσσια διάσταση των τέντη. Η αναθεώρηση των τέντη που θα γίνει ως ο Σονούπο θα είναι μια τεράστια ευκαιρία για να διαμορφώσουμε την θαλάσσια διάσταση των τέντη και θα πρέπει όλα αυτά να τα εντάξουμε σε ένα συνολικό πλαίσιο προς όφελος του Ευρωπαϊκού Θαλάσσιου Χώρου. Θα πρέπει να τονίσουμε την ε, διασύνδεση όλης της αλυσίδας μεταφορών, ε, η διασύνδεση των ε, λιμανιών, ας πούμε, που είναι στη θάλασσα και εκτός, πρέπει να είναι θέμα προτεραιότητας. Πρέπει να τα λάβουμε αυτά υπόψη μας ε, στις κατευθυντήρε γραμμές TNT. Θα πρέπει να γίνει, εδώ, εδώ ε, μάλλον εσείς οι Τραν θα έχετε μία έκθεση πρωτοβουλίας για αυτό το θέμα. Σας υποστηρίζω σε συνεδριάς που θα κάνουμε και για να ανταλλάξουμε απόψεις, ούτως ώστε να φτάσουμε σε κοινά συμπεράσματα. Προκειμένου να υπάρχει καλύτερη διασύνδεση των διαδρόμων πρέπει να δούμε, ε, να δούμε την ειδική διάσταση των ε, θαλάσσιων λεκανών. θα, υπάρχουν, ε, θα υπάρχει ένα πρόγραμμα εργασίας που θα παρουσιάσουν τα κράτη-μέλη για αυτό το θέμα τις επόμενες εβδομάδες. Επίσης, οργανώσαμε και κοινέ ομάδες εργασίας ανά λεκάνη με τους συναδέλφους μου από τους άλλους διαδρόμους. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πώς θα συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε και νέους προορισμούς ίσως. Οργάνωσα μία ομάδα εργασίας για τον Ατλαντικό μαζί με τους συναδέλφους που τους έχετε ακούσει τις τελευταίες εβδομάδες για το θέμα της διασυνδεσιμότητας των νησιών εν ώψη του Brexit. Αυτό το γεωπολιτικό θέμα είναι, δείχνει ξεκάθαρα το πώς θα λειτουργούν οι αυτοκινητόδρομοι αυτοί. Ε, ας πούμε, μπορεί να είναι μια εναλλακτική λύση, ε, ε ας πούμε η διασύνδεση νησιών με τη Γαλλία, ξέρω εγώ, στην, στους σημερινούς διαδρόμους μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, Πρέπει να δούμε τις προκλήσεις του θαλάσσιου τομέα και θα του δούμε χάρη στις αυτοκινητοδρόμους. Θα πρέπει να πρασινίσει ο θαλάσσιος τομέας και να υπάρξει ψηφιοποίηση ε, των ε, λιμανιών και, της, ε, και του κλάδου. Υπάρχουν 50 προγράμματα ύψους 436 εκατομμυρίων ευρώ που συνδέονται με το πρασίνισμα 1,6 δισεκατομμύρια χρηματοδότηση για θαλάσσιες μεταφορές, προγράμματα θαλασσίων μεταφορών, ε, ούτως ώστε να αλλάξει ο τρόπος που μεταφέρουμε εμπορεύματα και ανθρώπους. Πρότεινα τρεις θεματικούς πυλώνες στα κράτη-μέλη για το επόμενο πρόγραμμα. Πρώτον, ανάπτυξη α, βιώσιμων, ε, απρόσκοπτων και έξυπνων τέτοιων θαλασσίων χώρων. Καταρχάς, για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, να βελτιώσουμε τον αέρα και, την, το νερό, επενδύσεις για την απανθρακοποίηση και καινοτομία και οικολογικά κίνητρα. Δεύτερος πυλώνας. Θα πρέπει να έχουμε απρόσκοπτες θαλάσσιες μεταφορές, ε, να βελτιώσουμε την, ε, ε, τις πολύτροπες μεταφορές, ούτω ώστε να συνδεθούμε περισσότερο με τις περιφερειακές και απόμακρες περιοχές. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ένας έξυπνος θαλάσσιος ευρωπαϊκός χώρος με τη χρησιμοποίηση ε, ψηφιακών εργαλείων σε όλο τον κλάδο, με ψηφιοποίηση των, ε, της των συνδέσμων διαχείρισης της κυκλοφορίας. Ο στόχος μου είναι να δημιουργήσουμε μια ισχυρότερη θαλάσσια διάσταση των TEN-T που θα συνδέει ε, τα λιμάνια στην, που έχουμε στη θάλασσα με τα χερσαία τεντή. Έτσι θα έχουμε ε, καλύτερη ε, και πιο βιώσιμες μεταφορές ε, στη θάλασσα και στον, στην αυσιπλοεία. Η Πράσινη Συμφωνία είναι σημαντική για να υλοποιήσουμε τους στόχους για καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής Όμω δεν λάβαμε υπόψη μα την αυσιπλοεία στην Πράσινη Συμφωνία. Είναι κρίμα, γιατί είναι βιώσιμο ε, τρόπο μεταφορών. Αυτό είναι προβληματικό κατά την απόψή μου. Γιατί τα δύο πέμπτα του ε, ενδοενωσιακού εμπορίου ε, κατόγκο ε, μεταφέρεται μέσω της ναυσιπλοείας. Έχει τεράστιο δυναμικό, πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Θα ήθελα να υπάρχει ε, υποστήριξη από την Επιτροπή σας γι' αυτό θα σήμουν ευγνώμων για κάτι τέτοιο. Υπάρχει το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, που όμως δεν αναφέρεται σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Θα πρέπει να το συζητήσουμε. Και κλείνοντας, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ελπίζω να ακούσω πολλές ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος, για τα όσα μας είπατε. Και ευθύσαμε να δώσουμε τον ε, λόγο στον ε, κύριο Ρουέτε. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ και για πρώτη φορά να σας μιλήσω για αυτά τα οποία έκανα ως συντονιστής από τις αρχές του περασμένου έτους. Γνωρίζω ότι θα τα λέμε περισσότερο και όπως ο κύριος Μπόντεβεκ για ασχοληθεί με αυτή την έκθεση της πρωτοβουλίας για το ERTMS. Θα τα πούμε τον Μάιο και θα έχουμε την ευκαιρία επομένως να είμαστε σε επαφή. Κοιτάξτε τι έχω από το ERTMS, ότι αργήσαμε πολύ. Πάρα πολύ. Ταυτόχρονα όμως ε, πέρσι επιταχύναμε και αυτό είναι σαφές. Οπότε γι' αυτό σας λέω. Δεν είναι πλέον το ζήτημα του εάν θα ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση. Το θέμα είναι πότε και πώς. Οπότε με το δικό σας πολιτικό έλεγχο επιταχύνουμε το πότε, το δε, πώς θα απλουστευτεί. Μας πήρε πολύ χρόνο γιατί δεν υπήρχε το θεσμικό πλαίσιο. Είχαμε το συνδρομικό πακέτο, είχαμε την αρχή των συστημάτων, την ΙΝΕΑ, την ε, Τράπεζα Επενδύσεων και επίσης ε, τη στιβαρή διεύθυνση της DigiMove, οπότε μπορούμε να πούμε ότι για το ERTMS όλοι συντονισμένα προσπαθούμε. Και είμαι σχετικά σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε τελευταίο χρόνο με όλους τους εμπλεκομένους συνεργάζομαι κρατικές αρχές, ε, παρόχους, ε, ε, εταιρείες, ε, διαχειριστές υποδομών. Μην σας ε, πω τι έκανα μέρα προς μέρα πέρσι, αλλά είχα 90 συναντήσεις και μετά από αυτή την ενθουσιώδη εισαγωγή πάμε τώρα σε κάποια ομά στοιχεία. Έχουμε αυτό το σχέδιο ανάπτυξης του URTMS και βάζω μια ανωτελεία για να ε, επενέσω τον ε, Καρλ Βίνξ, τον ε, προκάτοχό μου, που τόσα χρόνια πάλεψε για να μείνει στο θεματολόγιο αυτή η υπόθεση. Έχουμε 15.000 χιλιόμετρα, μέχρι το 2030 πρέπει να καλυφθούν και έχουμε όπως βλέπετε εδώ, ε, σήμερα κάνει 5.800 χιλιόμετρα και ε, ακόμα είμαστε πίσω σε σχέση με το ERTMS ε, σε παγκόσμια κλίμακα και τώρα είμαστε στο 36-37% όσον αφορά την υλοποίηση με στόχο το 23. Πάρα πολύ σημαντική χρονιά αυτή γιατί έχουν υποσχεθεί τα κράτη-μέλη να γίνουν 40.000 χιλιόμετρα μέχρι το 20 και έχουν γίνει κάποιες καθυστερήσεις ήδη όσον αφορά τις προηγούμενες δεσμεύσεις αλλά είναι υποέλεγχο δεν λέω τίποτα άλλο πάμε τώρα σε ένα δεύτερο σημείο προβληματισμού κάτι που το παραβλέψαμε αρχικά θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρξει φιλόδοξο πρόγραμμα για ανανέωση και refitting των ατμομηχανών αλλά και των βαγονιών και των οχημάτων για τους διαδρόμους ε, για όλες τις χώρες και παντού 15.000 και έως έως 21.000 νέα οχήματα μέχρι το 2030, αλλά χρειάζεται να γίνει και κάποια προσαρμογή retrofitting 8500 13.000 άτομα μηχανών. Δύσκολα πράγματα, ψηλά ο πύχης, αν κάτσετε να σκεφτείτε τι κάνουμε ετησίως σε σχέση με το retrofitting. Οπότε έχουμε αυτή τη στρατηγική της ανάπτυξης της πολιτικής αυτής από οικονομικής δεν είναι λογικό. Εάν επιμερούμεθα μόνο τις υδροτροχίες και όχι τα οχήματα. Μιλάμε για δαπάνη 1,2 δις. Πριν είχαμε 2,9 για την προϋποδότηση του ERTMS, ακόμα έχουμε το Blending Facility και τώρα μπορούμε να το εφαρμόσουμε και σε πρωτότυπα, το ERTMS, άρα πολλά γίνονται για την χρηματοδότηση. Χρειάζονται όμως περισσότερα, αν θέλουμε να επιταχύνουμε το ρυθμό μας. πόροι από τα περιφερειακά ταμεία, εθνικοί πόροι, πόροι από την επενδυτική τράπεζα, την ΕΤΕ. Οπότε όλοι που ασχολούμεθα με το θέμα χρειαζόμαστε ένα σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης για να μπορέσουμε να εκμελευτούμε τις βιομηχανικές, τις τεχνικές δυνατότητες και μην έχουμε σκοτσέζι κοντούς. Γιατί ο χρόνος πιέζει. Πάντως, δύο άλλα σημεία προβληματισμού. Πρώτον, Έχουμε πάνω από 20 συστήματα σήμανσης ε, ε, όλα τα κράτη-μέλη. Άρα πρέπει να πάμε σε βαθμία κατάργηση. Και θέλουμε αυτά να τα συζητήσουμε τις επόμενες μήνες. Να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτή η βαθμία κατάργηση αυτών των συστημάτων β' κατηγορίας. Γιατί μας πήρε τόσο καιρό γιατί οργανώνουμε την μετάβαση από το παλιό στο νέο. Η μετάβαση είναι όλο ένα πιο περίπλοκη και όλο ένα πιο δαπανηρή εάν θα πρέπει συνέχεια να μπερδευόμαστε με το παλιό σύστημα. Ένα αυτό. Το δεύτερο πρέπει το ERTMS να απλωστευθεί. και να καταλάβουμε ότι μιλούμε για ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης του σιδηροδρόμου και όχι μόνο για σηματοδότηση και τέτοια. Είναι καινούργια πράγματα, άρα πρέπει να οργανωθούμε με έναν τρόπο οργανωμένο και όχι σπασμωδικό για το μελλοντικό ERTMS. Ολοκληρωμένο και συνεπή συνεχή. Τώρα, γιατί την τελευταία εμπειρία, η εμπειρία μου ήταν ότι όπου και ό,τι να λέγανε για το ERDMS είναι αποδεικτό ότι πρόκειται για τον χρυσού κανόνα, για την πανάκια. Άρα θα πρέπει να οργανώσουμε αυτήν την περίπλοκη μετάβαση. Και αν το κάνουμε ταχαίως, τότε θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να έχουμε πιο αποτελεσματικούς στυροδρόμους. Και συμφωνώ με αυτά που είπατε για την ε, ναυσιπλοεία. Αλλά βιώσιμες μεταφορές πάνω πει σιδηρόδρομος, άρα εκεί δίνουμε τη μάχη. Ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας δεν χάνουμε χρόνο. Θα δώσω το λόγο κατευθείαν στο συντονιστέ. Ο κύριος Μαρινέσκου, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, και χαίρομαι που σας βλέπω ξανά. Κύριε Μπόντιβικ. Ευχαριστώ τον κύριο Ετιέν που με αντικατέστησε σήμερα το πρωί. Άκουσα πολύ καλά σχόλια για την προεδρία του. Κύριε Μποδεβίκ, μιλήσατε για την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα της ναυτιλίας, αλλά δεν άκουσα κάτι συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν ε, μπορείτε να μας, ε, διαφωνεί, μας διαφωτίσετε. Και δεν ξέρω αν έχετε αξιολογήσει ένα σύστημα ferryboat για να μεταφέρουν φορτηγά από την Τουρκία, στην Ιταλία, ξέρω εγώ, στη Βενετία, στη Γένο, για να μειωθούν οι εκπομπέ. Ε, για τις οποίες μιλάμε. Και κύριε Ρόιτ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνετε. Το RTMS είναι ένα πολύ καλό σύστημα αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή. Εάν έχετε λάβει υπόψη την κατάσταση της διαλειτουργικότητας, ε, ενορμόνησης και τυποποίησης των σιδηροδρόμων, αλλά και για το ERTMS ε, η διαλειτουργικότητα, έχω διαβάσει, ότι δεν είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές των συστημάτων, κάτι το οποίο δεν χρειαζόμαστε. Και ξανά, Green Deal. Μεγάλη συζήτηση, το ξέρω. Μετακίνηση στον σιδηρόδρομο. για τους διαδρόμους ε, τώρα φορτίων που δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή όπως είχε προβλεφθεί πριν από 7-8 χρόνια. σκοπεύετε να εφαρμόσετε το ERTMS σε όλους τους διαδρόμους. Στα αλήθεια όμως, να είναι τα πάντα διαλειτουργικά για να είναι ελκυστικά για τις εταιρείε να μεταφέρουν έτσι τα αγαθά. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντάνιελσον για τους σοσιαλιστές. Ε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για τις παρουσιάσεις σας. Όσον αφορά τους αυτοκινητοδρόμους της θάλασσας, έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, πού βρίσκονται οι στενοποί αυτή τη στιγμή ε, όσον αφορά την υλοποίηση των έργων. Μετά. Δεύτερον, μιλήσατε για το ότι ο πρώτος πυλώνας πρέπει να είναι η βιωσιμότητα σύμφωνα με τις φιλοδοξίε κομισιών ε, κτλ. Αλλά συγκεκριμένα, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις ε, για να γίνει ο τομέας της ναυτιλίας πιο βιώσιμος. Και τρίτον, όσον αφορά την διαλειτουργικότητα, γιατί εδώ πέρα συμφωνώ ότι πρέπει να λυθεί αυτό, έχετε κάποια συγκεκριμένα καλά παραδείγματα τα οποία θα θέλατε να μας παρουσιάσετε κάποιες χώρες, ε, περιφέρειες όπου υπάρχει ακριβώς, ε, υπάρχουν αυτές οι συνδυασμένες μεταφορές. Μετά, σε σχέση με το ERTMS. Όπως είπε και ο κύριος Μαρινέσκου, είναι ένα σύστημα κλειδί για να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί σωστά στην Ευρώπη. Βγήκα ε, κάποια στιγμή, δεν άκουσα ολόκληρες τις ομιλίες σας, αλλά ακόμα και αν αυξάνεται ο ρυθμός, ε, ξεκολουθούμε να ε, είμαστε, να υστερούμε λίγο. Και έχω την εντύπωση ότι το σύστημα γίνεται όλο και πιο επίμαχο, γιατί έχουμε περιφέρειες όπου τώρα αρχίζει να αναπτύσσεται και έχει κάποιο κόστος και μέχρι να γίνει ένα πραγματικά πανευρωπαϊκό σύστημα μπορεί κάποιος λογικά να αμφισβητήσει την σκοπιμότητα του να επενδύει πολλά λεφτά σε ένα τοπικό σύστημα. Δηλαδή κάποια στιγμή θα υπάρξει ένα σημείο καμπής όπου δεν μπορεί πλέον να δικαιολογήσει πολιτικά δαπάνες σε ένα άλλο σύστημα. Ρεαλιστικά πότε το βλέπετε να συμβαίνει αυτό. Γιατί βεβαίω και οι περιφέρειε μετά σκέφτονται γιατί να το κάνουμε εμεί αν όλο το σύστημα έχει μείνει πίσω. Ευχαριστώ. Κύριε Ρικέ, έχετε τον λόγο. Content de revoir euh, Χαίρομαι που βλέπω εδώ τους συντονιστές ξανά. Μία ερώτηση. Στις, στους θαλάσσιους αυτοκινητοδρόμους μπορούμε να βάλουμε και τον τομέα της α, ναυσιπλοείας, της μεταφοράς φορτίων, δηλαδή διαθαλάσσης. <coughs> Γιατί στα πλαίσια του Brexit θα θέλαμε κάτι τέτοιο γιατί θα μας εξασφαλίσει απρόσκοπτες μεταφορές. Κύριε Ρούτε, ένα οικονομικό ερώτημα. Ποιος και πώς ε, χρηματοδοτεί ε, το υλικό που μεταφέρεται μέσω του ERTMS. Έχουμε πιστώσεις συγκεκριμένες. Οι μεταφορικές εταιρείες το χρηματοδοτούν συνδέεται με τις ε, πιστώσεις των, ε, για τις επενδύσεις. Δεδομένου του όγκου ε, της σημασίας αυτής, ε, ανησυχώ για το ποιος κάνει τη χρηματοδότηση. Ο κύριος Καφ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Να αναφερθώ και εγώ σε ερώτηση του συναδέλφου για την χρηματοδότηση. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα περισσότερα για το ποιος θα πληρώσει για το ETRMS. Και όσον αφορά τώρα τα προβλήματα που υπάρχουν και την αργή ανάπτυξη του συστήματος, μπορούμε να κατηγορήσουμε περισσότερο τις εταιρείες ή τις χώρες που βρίσκονται τα εμπόδια. Εμφανίζονται στο επίπεδο σιδηροδρομικών εταιριών που δεν θέλουν αυτήν την τεχνολογία είναι πρόβλημα απλώς ε, των εθνικών, ε, στο εθνικό επίπεδο. τα ήθελα της απόψεις σας. Και μετά όσον αφορά τα ζητήματα της ε, ναυτιλίας. Είδα αυτά τα οποία αναφέρατε ως προκλήσεις για την Ιρλανδική νήσο και το Ιρλανδικό κράτος μετά από το Brexit. Θα μπορούσατε ίσως να επεκταθείτε. Γνωρίζω πως ε, έχουν συζητηθεί επιπλέον δρομολόγια φεριμπότ μεταξύ της Νότιας Ιρλανδίας και της Γαλλίας ε, ή της ε, Ολλανδίας ή άλλων λιμένων. Και θα ήθελα κάποιο σχόλιο για την αυσιπλοεία μικρών αποστάσεων και τι ρόλο μπορεί να παίξει. Και αν υπάρχει κάποιος ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις υποδομές ε, των λιμένων για να δοθεί ένα επιπλέον κίνητρο για τα μικρά αυτά δρομολόγια. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για δύο λεφτά. Δεν θα μιλήσω αγγλικά εγώ, λέει ο κύριος Κάμπο Μενόζη. Προς τον κύριο Ρούτε. Θα μιλήσω αγγλικά. Λοιπόν, είπατε ότι σκοπεύετε να βελτιωθεί το σύστημα ERTMS Μιλήσετε για 100 εκατομμύρια ευρώ και τη σχετική ψηφιοποίηση. Ε, είναι δύσκολο να πετύχουμε τον στόχο του 2030. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να υπάρξει η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να δοθούν περισσότερα χρήματα στο ERTMS, ίσως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κτλ αλλά αυτή τη στιγμή λίγο πολύ έχουμε μια κάλυψη 10%. Τα δεδομένα σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ε, θεωρείτε ότι θα πάει προς αυτή την κατεύθυνση η Κομισιόν για να τα σεβαστεί αυτά. είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για ένα ευρωπαϊκό μοντέλο. Ευχαριστώ, Φιντέσα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε και εσείς κύριε Ρουτ. Είχαμε γνωριστεί πριν από πολλά χρόνια επικεφαλής της ε, Digimove. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Μπόντεβικ, δεν άκουσα την παρέμβασή σας, δεν θα κάνω ερωτήσεις. Θα επικεντρωθώ στο ERTMS. Μας ανησυχεί ε, το ότι δεν υπάρχει πρόοδος και ακριβώς ε, σωστή είναι αυτή η έκκληση για να βρεθούν περισσότεροι πόροι, αλλά μέχρι στιγμής δεν εισακούγεται. Οπότε θα έπρεπε να υπάρξει ένας ε, συνδυασμός διαφόρων πηγών χρηματοδότησης. Το μέσο συνδέοντας στην Ευρώπη, το InvestEU, ε, να υπάρξει ένα συνδυασμός και με εθνικές ε, χρηματοδοτήσεις για να έχουμε ένα φαινόμενο μόχλευσης για να κινητοποιηθούν και ιδιωτικές ε, επενδύσεις. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω σε ποιο σημείο έχει φτάσει ο διάλογος με την Κομισιόν για αυτήν την πρόταση που νομίζω περιγράψατε κι εσείς. Και νομίζω είναι σαφές σε όλους το πόσο μπορεί να ωφελήσει το Green Deal ε, το σύστημα αυτό το ERTMS γιατί ε, πολλά λέγονται αλλά η εφαρμογή μιας τέτοιας ε, τεχνολογίας θα μας έδινε την δυνατότητα να εντείνει η πυκνότητα των ε, δρομολογίων χωρίς νέες υποδομές. Προφανώς έτσι λοιπόν θα είχαμε μετακίνηση των φορτίων στο σιδηρόδρομο, μείωση των εκπομπών κτλ. Οπότε νομίζω αν υπάρξει και η κατάλληλη πολιτική στήριξη θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τους σχετικούς πόρους. Ευχαριστώ κυρία Κουντουρά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, να ευχαριστήσω τον κύριο Μπόντουικ για την τοποθέτησή του. Το νέο Green Deal που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να μειώσει τις εκπομπές από τις μεταφορές κατά 90% και για να το πετύχει αυτό θέτει ως προτεραιότητα να μειώσει σημαντικά το ποσοστό των οδικών μεταφορών που σήμερα βρίσκεται στο 75% των συνολικών μεταφορών αυξάνοντας το ποσοστό των σιδηροδρομικών μεταφορών και την εσωτερική ναυτιλία στους ποταμούς από τη στρατηγική αυτή για την αλλαγή του μείγματος μέσων μεταφοράς, όπως και εσείς επισημάνατε, απουσιάζει η παραδοσιακή θαλάσσια ναυτιλία μικρών αποστάσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με την Επιτροπή, τα δύο πέμπτα των ενδοκινοτικών ανταλλαγών πραγματοποιείται μέσω της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων, από την οποία εξαρτάται αποκλειστικά, όπως γνωρίζουμε, και η νησιωτικότητα έχετε εργαστεί για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της θαλάσσιας ναυτιλίας μικρών αποστάσεων μέσω του ΝΤΕΤΗ. Ζητήσατε τη βοήθειά μας και βεβαίως θα την προσφέρουμε. Γι' αυτό θα ήθελα να, ε, την άποψή σας για το ρόλο που μπορεί να παίξει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Green Deal κάποιες ε, πληροφορίες ώστε να ενημερωθούν και οι συνάδελφοι. Επίσης, καθώς οι λιμένες αποτελούν εμπορικές πύλες όχι μόνο του κράτους μέλους το οποίο βρίσκονται, αλλά έχουν σαφώς διεθνή χαρακτήρα, ίσως θα έπρεπε να έχουν και στήριξη ως διασυνοριακά έργα. Θα ήθελα την εποψή σας και σε αυτό. Τέλος, προτείνω να έχουμε μία επαφή και με τους υπόλοιπους σκιώδεις εισηγητές, ώστε να συνδιαμορφώσουμε προτάσεις για την αναθεώρηση του ΤΕΝΤΗ, γιατί όπως βλέπουμε υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Merci beaucoup. Allez, nous continuons. Désormais... Συνεχίζουμε. Η κυρία Μπιλμπάου, ένα λεπτό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ρούτε, έχουμε θετικά νέα, νέα. Προχωράμε, επιταχύνουμε μάλιστα. Όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω ότι λέτε πως έχουμε ελεγχόμενες καθυστερήσεις. Τι εννοείτε ακριβώς. Επίσης, έχουμε 20 συστήματα σηματοδότηση σήμανση. Πώς θα τα μειώσετε. Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων εδώ μεταξύ των, ε, χωρών. Έχετε μια στρατηγική για να μειώσετε αυτά τα διαφορετικά συστήματα ε, κατηγορίας Β και μέχρι πού μπορούμε να προχωρήσουμε. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε επαρκή μετάβαση και να φτάσουμε σε ένα ανταγωνιστικό σύστημα και πιο βιώσιμο εάν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην οικοδόμηση, στην υλοποίηση των TNT. Μπορούμε να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα επίπεδα χωρίς να προχωρήσουμε στο TNT. Τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για να πείσουμε τα κράτη-μέλη να ολοκληρώσουν αυτά τα προγράμματα και να τα πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι αυτά είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη, αυτά τα προγράμματα. Η κυρία Γκραμπίνη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Γκραπίνη. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Ο πρώτος μας ομιλητής. Είπατε για ένα ευφυές σύστημα θελήσεων μεταφορών και είπατε ότι ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα των ε, λιμμένων και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το ERTMS σχετικά με αυτό, γιατί μας είπατε ότι θα γίνει, δεν μας είπατε όμως το πότε. Μερικοί λένε ότι έχουμε 20 συστήματα ε, σηματοδότησης διαφορετικά, έχετε κάποιο προγνωστικό. Πότε αυτό θα έρθει εις πέρας επίσης για την διαλειτουργικότητα και την συνδεσιμότητα τι θα γίνει, μια που υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα. Πότε θα φτάσουμε στο σωστό επίπεδο, δεν χρειάζονται επενδύσεις σε υποδομές. Πέστε μας μερικά στοιχεία. Πες μας θα γίνει με αυτό το όριο, το στόχο χιλιόμετρων 2 το 2020, θα τα έχουμε καταφέρει μέχρι τότε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκραπίνη. Εσείς κύριε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Καλτσκίν. Μας είπατε ότι η αυτοκινητόδρομη της θάλασσας πρέπει να ευθυγραμμιστεί μάλλον με το κεντρικό δίκτυο και τους σχετικούς διαδρόμους και είπατε επίσης ότι θα πρέπει να προσεχθεί περισσότερο η περιφέρεια. Εγώ προέρχομαι από μια περιφέρεια, από μια πόλη της περιφέρειας, την Μπρέστ. Είμαστε μόνοι πόλοι πάνω από 100.000 που είναι τόσο απομακρυσμένοι από οποιοδήποτε διάδρομο του κεντρικού δικτύου. Κοίταξε το χάρτι. Δεν ξέρω, μπας και αυτό ισχύει και για το βορρά της Σουηδίας, δεν ξέρω. Εντάξει, από πλευράς χωριού μου το βλέπω αυτό, αλλά το ίδιο το βλέπουν και οι ψηφοφόροι μου. Τι θα κάνετε, πώς θα μπορέσετε να καλύψετε την περιφέρεια. Δεν θα το μπορέσετε αν ευθυγραμμιστείτε και προσέξετε το κεντρικό δίκαιο. Η πρόεδρε, σε ευχαριστούμε. Βίντε. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Να σας τα πω στα δανέζικα. Αυτές οι διευκολύνσεις όπως λέμε χρειάζονται. Για να υπάρξει ισορροπία μεταξύ χερσιών μεταφορών, σιδρομών, θαλασσίων. Θα πρέπει να γίνει αυτή η ευθυγράμμιση και η ισορροπία σε πολλά μέρη. Ένα λεπτό έχετε και εσείς το λόγο. Κυρία. Ναι, καλημέρα κύριε Μπούτεβη, κύριε Ρούτε, καλημέρα και σας ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσει. Η πρώτη είναι πώς θα διασφαλίσουμε ότι οι χώρες ε, που έχουν προχωρήσει μπροστά με το ERTMS δεν θα μείνουν πίσω όταν περάσουμε στην στήριξη γιατί ε, Κάποιοι σκέφτονται ότι ας μην κάνουμε τίποτα μέχρι να το χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κρίμα τελικά αυτό να είναι μειονέκτημα για αυτούς που προχωράνε μπροστά. Και το δεύτερο ερώτημα είναι η σχέση μεταξύ των δύο έργων που θα λειτουργήσουν καλύτερα αν συνεργάζονται. Πώς ε, θα τα καταφέρουμε να έχουμε ένα έξυπνο δίκτυο σιδηροδρόμων που θα έχει και τη σύνδεση με την θάλασσα. Πώς ε, σκοπεύετε να συνδέσετε τα δύο δίκτυα. Σας ευχαριστούμε κυρία Ντεπαρνέ. Τώρα η σειρά μου. Έχω δύο μεγάλα ερωτήματα. Μα μιλήσατε για την Πράσινη Συμφωνία. Τι περιμένετε από την Πράσινη Συμφωνία και ποιε είναι οι συγκεκριμένε προτάσει σα για το τι πρέπει να περιέχει η Πράσινη Συμφωνία. Δεύτερο σημαντικό κατ' με, είναι ότι μα μιλάνε για του θαλάσσιου αυτοκινητοδρόμου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 20 χρόνια. Παράλληλα, υπάρχει Υπάρχουν διάφορες λύσεις. Ε, το G20 μας λέει ότι για το θαλάσσιο τομέα θα πρέπει να μειώσουμε τις θαλάσσιες μεταφορές. Και από την άλλη εμείς θέλουμε να φτιάξουμε τους θαλάσσιους αυτοκινητοδρόμους. Ε, συμφωνήστε. Αν θέλουμε τους αυτοκινητοδρόμους, τους θαλάσσιους αυτούς, πρέπει να τους τελειώσουμε. Πώς θα πείσετε τα κράτη-μέλη και θα τα θέσετε ενώπιον των ευθυνών τους. Επίσης, για το τρένο, για το σιδηρόδρομο. Χθε ε, εγκαινιάσαμε νέο αυτοκινητόδρομο προς τις Βρυξέλλες, ε, το νυχτερινό τρένο που φτάνει στις Βρυξέλλες. Ε, εδώ μας ενδιαφέρουν οι πολύτροπες, συνδυασμένε μεταφορές. Τι θα κάνουμε στα λιμάνια, ε, τα οποία θα πρέπει ε, να συνδέονται, να έχουν δηλαδή ε, κέντρα, ούτως ώστε από τα λιμάνια να πηγαίνουμε κατευθείαν στο σιδηρόδρομο. Ε, πολλά λιμάνια έχουν τέτοιες συνδρομικές ε, μεταφορές, αλλά πώ μπορούμε να τα συνδυάσουμε πραγματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα δύο. Έχετε πέντε λεπτά για να απαντήσετε σε όλε αυτέ τις ερωτήσεις. Δεν είναι εύκολο, το ξέρω, αλλά έχουμε πολύ μετρημένο χρόνο. Ο κύριο Ροντίκ, πρώτος και καλύτερος. Να απαντήσω τότε στα γερμανικά. Να απαντήσω πρώτα απ' όλα που είναι τα ελλείμματα. Ε, υπάρχουν διάφορα. Υπάρχουν λιμάνια ακόμα στην Ευρώπη τα οποία δεν έχουν συνδυασμένες ε, μεταφορές. Δεν έχουν παραδείγματος χάρη σιδηροδρομική σύνδεση. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο εστιάζουμε. Ταυτόχρονα από την άλλη πλευρά έχουμε ένα προβληματικό σύστημα για την φόρτωση. Οπότε θα θέλαμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα το οποίο παραδείγματος χάρη θα αφορούσε τις τελωνιακές διατυπώσεις. Επίσης έχουμε την ε, διαχείριση της κίνησης ε, στην ε, θάλασσα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Βαλένθια και η Βαρκελόνη έχουν μια σύνδεση με την Τσίβιτα Βέκιο που συνεχίζει μετά προς Αγκώνα και μέσω της Αδριατικής προς Κροατία, Σλοβενία, η Δυτικά Βαλκάνια μέχρι την Ελλάδα. Αυτό ε, επιτυγχάνει πάρα πολλές ε, μειώσεις των εκπομπών, μειώνει κατά πολύ το χερσαίο δρομολόγιο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε δηλαδή, ε, είναι κάτι το λειτουργεί και αν δούμε στα σοβαρά το Green Deal θα μπορούσαμε το 2050 να έχουμε πλοία με υδρογόνο να κάνουν αυτά τα δρομολόγια και να πετύχουν τους στόχους που θέλει η Κομισιόν και η Κοινοβούλιο. Βεβαίω αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε λεφτά. Έχουμε διάφορα στον τομέα της έρευνας ε, που πρέπει να αναπτυχθούν. Μπορούμε λοιπόν να πετύχουμε πολλά με νέες ιδέες. Το δεύτερο είναι τα λιμάνια που αναφέρθηκαν. Εδώ πέρα πηγαίνει η ψηφιοποίηση. Πρέπει να μειωθούν οι γραφειοκρατικές ε, διατυπώσεις, αλλά βεβαίως πρέπει να είναι προστατευμένες και από πλευράς ασφαλείας οι λιμενικές εγκαταστάσεις, οπότε μπορεί εδώ πέρα η ψηφιοποίηση να μας βοηθήσει πάρα πολύ. Θα ήθελα ταυτόχρονα να πω ότι αν θέλουμε να δώσουμε κίνητρα, συζητάμε για θετικά κίνητρα, το οικολογικό μπόνους στην Ισπανία, στην Ιταλία, το απόγευμα έχουμε και μια σχετική συνάντηση, όπου προσπαθούμε ακριβώς να δούμε πώς θα επιβραβεύσουμε αυτούς που αντί για 5.000 χιλιόμετρα με το φορτηγό τα βάζουν ε, σε, μια, σε ένα πλοίο και κάνουν ένα μικρό ναυτικό δρομολόγιο. Ένα άλλο ερώτημα. Αναφερθήκατε βεβαίως ε, εσείς ε, και στα λιμάνια τα οποία σας απασχολούν ε, στις περιοχές σας κατανοητό. Δεν είναι πάντα ως κάτι το εναλλακτικό. Μπορούμε να έχουμε ακριβώς ε, την ανάγκη για αυτά τα λιμάνια, για τις απομακρυσμένες περιοχές, για την γειτονία. Ε, στην Αφρική παραδείγματο χάρη, όπου βρισκόταν η τα τελευταία χρόνια η χώρα με την δεύτερο μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης. Μπορούμε λοιπόν να μετατοπίσουμε ακριβώς ε, τις συγκοινωνίες απευθείας στη θάλασσα. Προς τον κύριο Ντάνιλσεν μια απάντηση τι είναι τελικά αυτή η περιφέρεια η οποία λειτουργεί. Αν μπορούμε να δούμε π.χ. την Βαλτική. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με έντονη κίνηση σε σημείο που σκεφτόμαστε ε, να δούμε πώς ε, θα γίνει καλύτερη για να μεταφερθεί ακόμα μεγαλύτερος όγκος ε, εκεί πέρα. Υπάρχουν όμως προβλήματα που μπορώ να σας παρουσιάσω. Υπάρχει εξή κατάσταση στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε κάτι εάν συνδέουμε ένα βασικό λιμάνι με ένα συμπληρωματικό λιμάνι. Γιατί λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε στην αναθεώρηση πως συνδέσουμε δύο συμπληρωματικά λιμάνια εάν με αυτόν τον τρόπο μετατοπίζεται η κίνηση από τους δρόμους στη θάλασσα. Και τελευταίο, τι μπορεί να γίνει για τη συνεργασία μεταξύ σιδηροδρόμων και ναυτιλίας μικρών αποστάσεων. Αυτό οφείλεται, αυτό βεβαίως πρέπει να πάει στην υπεραιτέρω ανάπτυξη των λιμανιών, αλλά και μια τελείως διαφορετική εφοδιαστική αλυσίδα γιατί ε, κατά κανόνα κυρίαρχος είναι ο δρόμος εδώ πέρα. Αν τα καταφέρουμε αυτά θα επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο και αν παίρνουμε στα σοβαρά τον Green Deal θα πρέπει πραγματικά να συμπεριληφθεί και η ναυτιλία μικρών αποστάσεων. Και χαίρομαι βεβαίω να ξανάρθω στην Επιτροπή σας ε, να συζητήσουμε αυτά τα θέματα όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ. Έχετε τον λόγο και εσείς ε, για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να απαντήσω για κάποια θέματα που έθεσε ο κ. Μαρινέσκου για τη διαλειτουργικότητα, αλλά και άλλοι ευρωβουλευτές. Νομίζω ότι τώρα έχουμε μια διαφορετική κατάσταση από αυτή που είχαμε τις προηγούμενες δεκαετίες, τα προηγούμενα χρόνια. Ησυχία. Θα ακούσουμε τον ομιλητή μας ή όχι. Έχουμε μία αρχή για το σιδηρόδρομο, τη Βαλανσιέν, που είναι η αρχή που διαχειρίζεται το ERTMS και ρυθμίζει όλα τα προβλήματα διαλειτουργικότητας ε, που είχαμε στο παρελθόν και που τονίσατε. Η έγκριση για τη θέση στην αγορά περνάει από την αίρα η άγκριση για τις δημόσιες προμήθειες του RTMS περνάει από την ΕΡΑ, επομένως έχουμε ένα πρόβλημα ε, που είχαμε εντοπίσει. Δεν έχουμε πια το πρόβλημα που είχαμε εντοπίσει στο παρελθόν. Χρειάστηκε χρόνος για να το λύσουμε. Ο κ. Ντάνιλσον και ο κ. Μαρινέσκου ε, μίλησαν για του ελεύθερου διαδρόμους. Όταν αναπτύξουμε τους διαδρόμους φορτίου και συνδεθούμε με τα 10T ε, θα πρέπει να σκεφτούμε για τα δύο συστήματα παράλληλα και να τα αναπτύξουμε παράλληλα. Ε, στην επόμενη αναθεώρηση των 10T θα πρέπει ε, να δούμε μαζί τους διαδρόμους φορτίου μαζί με τα 10T. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουν περισσότερη στοιχεία λειτουργικότητας οι διάδρομοι αλλά οι διάδρομοι φορτίου χρειάζονται το ERTMS ε, για να γίνεται σωστά η διαχείριση του φορτίου, των εμπορευμάτων. Κύριε Ντάνιελσον. Έχουμε διάφορες περιφέρειες που εφαρμόζουν το ERTMS και ε, υπάρχουν κάποιες άλλες που δεν το κάνουν. Θα πρέπει να υπάρξει πλήρης εφαρμογή του ERTMS και να έχουμε και την απαραίτητη χρηματοδότηση βέβαια γι' αυτό. Κύριε Ρικέ, πολύ σωστά θέσατε το πρόβλημα του φορτίου το οποίο ε, μεταφέρεται δια θαλάσσης. Χρειάζεται μια στρατηγική ευρωπαϊκή. χρηματοδοτούμε ήδη μέσα στο ΣΕΦ αυτό το φορτίο. Αλλά υπάρχουν διαφορετικές στάσεις στα διαφορετικά κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την χρησιμοποίηση δημοσίου χρήματος, τη δημόσια χρηματοδότηση. Στην Ολλανδία, Φερρυπίν, έχουμε κάτι τέτοιο, το έχουμε και στο Βέλγιο, αλλά όχι κατά ανάγκη στη Σουηδία ή σε άλλες χώρες. Μερικές φορές με ψευδή επιχειρήματα. Ότι είναι δηλαδή κρατικέ ενισχύσει κάτι τέτοιο και αν δεν πρέπει να το κάνουμε. Αυτά τα επιχειρήματα πρέπει να τα ανασκευάσουμε. Και στο πρόγραμμα εργασία ε, που θα έρθει το Μάιο θα απαντάω σε αυτά τα θέματα, θα, θα σχολιάζω αυτά τα θέματα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ε, ερωτήσεις. Κυρία Μπιλμπά όμως, θέσατε ένα ερώτημα που είναι πολύ δύσκολο να επιλύσουμε. Πώς θα καταφέρουμε να υπάρχει υποχρέωση από τα κράτη-μέλη να σταματήσουν το σύστημα της κλάσης P. Και στη συζήτηση για τα T για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, αλλά και για το TSI SSS, πρέπει να σκεφτούμε ούτως ώστε να έχουμε μία ημερομηνία για να σταματήσει το σύστημα κλάσης P, τάξης P. Θα είναι πολύ δύσκολο, θα πρέπει να βρούμε λύσεις στις ε, δευτερογενείς ε, γραμμές, αλλά πρέπει να το καταφέρουμε, γιατί αλλιώς πάτε σε οποιαδήποτε γραμμή παραγωγής ε, για, τις, για τους υδροδρόμους και εκ των προσαρμογής. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το πράγμα, πρέπει να ε, υπάρξει επιτάχυνση. Για τη χρηματοδότηση να πω δύο λόγια και θα σταματήσω μετά. Πρέπει να κινητοποιήσουμε διαφορετικές ε, χρηματοδοτικές δυνατότητες. Έχουμε μια δυσκολία. Ποιος θα κερδίσει περισσότερο. Είναι ο διαχειριστής των ε, υποδομών αλλά ο διαχειριστής υποδομών δεν μπορεί ε, με βάση όλες τις νομοθεσίες να δώσει τα λεφτά στο, στους διοδρόμους. Ή θα ανέβουμε λοιπόν στον Υπουργό Χρηματο, ε, Οικονομικών και αυτός ας πούμε το ε, τη χρηματοδότηση γιατί εκ των υστέρων προσαρμογή είναι πάρα πολύ ε, σημαντική για το οικονομικό κέρδος ή θα βρούμε άλλες λύσεις είτε με ενωσιακά κονδύλια είτε με εταιρικέ σχέσεις δημοσίου ιδιωτικού ή με δυνατότητα συνδυασμενη χρηματοδοτηση Το Ιταλικό παράδειγμα είναι ενδιαφέρον. Ο Ιταλ... Ιταλική σιδηρόδρομοι έκανα μια καταπληκτική μελέτη και είδαν ότι είναι πολύ πιο φθηνό να υπάρχει το ERTMS. Αν το ενσωματώσετε στις υποδομές και δεν έχετε όμως τις, α, τις σειροτροχιές, ε, αν δεν έχετε τις ατμομηχανές είναι Ακριβώς. Και ίσως θα πρέπει να απομακρυνθούμε από την, ε, το, το χρονικό ορίζοντα του 2050. Να το κάνουμε πιο νωρί. Όχι μόνο να εφαρμόσουμε το ERTMS στου διαδρόμου, αλλά όπω κάνουν κάποια κράτη-μέλη. Σουηδία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ιταλία, Ιταλία το σκέφτεται, η Γερμανία το σκέφτεται. Να εφαρμόσουμε το ERTMS στο ουσιαστικό τμήμα του δικτύου, σε όλο το δίκτυο. Σας ευχαριστούμε. Θα είμαστε σε επαφή. Πρόκειται για δύο θέματα που μας ενδιαφέρουν, αλλά έχουμε δύο ερωτήσεις που είπε ότι κάποιες βίλες, κάποιες περιοχές που έχουν προβλήματα. Θα πρέπει να το δούμε αυτό και για το Πράσινο Σύμφωνο. Τι προσδοκάτε, πώς θα προχωρήσουμε, σιδηρόδρομοι, θαλασσίες μεταφορές, βέβαια να υπάρξει κινητοποίηση, είναι σημαντική και η χρηματοδότηση. Ευχαριστούμε που ήρθατε πάντα ευπρόσδεκτοι εδώ. Χειροκροτήματα για σας. Merci <laughs> <laughs> Allez, nous continuons nos travaux. Συνεχίζουμε, λέει Πρόεδρος. Allez, nous continuons. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, οι Ρωμανοί διερμηνείς, μπορείτε να μου κάνετε μία χάρη γιατί υπάρχει κάποια αντανάκλαση στο παραθυρό σας και μου έρχεται εδώ η αντανάκλαση του ηλίου στα μάτια. Αν μπορείτε να κατεβάσετε την κουρτίνα, τι έχετε εκεί. Eh ben regardez, les Roumains, ils ont pas de lucarne, mais ils ont mis une feuille pour leur présidente. Δεν έχουν κουρτίνα, αλλά τουλάχιστον βάλανε ε, αυτό το κομμάτι χαρτί για να σώσουν την πρόεδρο. Α, και, Α, και από τη γαλλική καμπίνα. Να τη, η προβληματική. Τέλος πάντων. Συμμορφώθηκαν οι Ρουμάνοι και σας ευχαριστούμε. Κύριε Μαρινέσκου, είπαμε, υπάρχει ένα παραθυράκι στο, στην καμπίνα των δερμηνέων και ακούω να μου λένε από τα ακουστικά οι δερμηνείς, δεν γίνεται αυτό ε, κυρία Αντελή, να βάλουν κάτι, μια που δεν υπάρχει, η, μια που δεν υπάρχει ε, κάποιο είδου παντζούρι ή κουρτίνα. Πάντα, πάντα οι Ρουμανοί βρίσκουν τις λύσεις, λέει ο κύριος Μαρινέσκου. Είναι απαραίτητο, απαραίτητο για την άνεσή σας. Α, σωστά. Πολύ ωραία. Οπότε, ξεκινάμε με το δεξί για της περίπτωσης ψηφοφορίας. Είναι μερικοί που σας βλέπω πρώτη φορά φέτος. Σας βλέπω τώρα πρώτη φορά, άρα καλή χρονιά σε εσά, την οικογένειά σας. Καλή επιτυχία, υγεία. Κύριε Γκραπίνη, καλά θα βιάζει να ψηφίσετε, αλλά εγώ επειδή είμαι ευγενική πρώτα σας εύχομαι. Άρα μια παραγωγική χρονιά, κυρίως εδώ στην Επιτροπή μας να κάνουμε μια δοκιμή, πριν ψηφίσουμε. Να δούμε και αν έχουμε απαρτία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Allez. Voilà, le vote est ouvert. Allez, je ferme le vote. Ψηφίζουμε, πέρας. Πολύ καλά. Δεν περισσεύουν ούτε σοσιαλιστέ, ούτε ΕΛΚ, ούτε τίποτα. Τα νούμερα βγήκανε. Οπότε, πρέπει να σας πω όμως ότι έχουμε τέσσερις ε, για επιβεβαίωση, για κάποιες συμφωνίες μετά από τη δεύτερη ανάγνωση. Απλή πλειοψηφία. Και θα γίνει ο διαδικασία μετά τις ψηφοφορίες Πρόκειται να απευθύνω επιστολή στον ε, πρόεδρο της Κορεπέρ και μετά το Συμβούλιο πρόκειται να προσαρμόσει τα της πρώτης ανάγνωσης και μετά θα διαβιαστεί ο φάκελος για τη δεύτερη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο. Και έτσι γνωρίζετε τώρα όλη τη διαδικασία. Προχωρούμε τώρα στην ψηφοφορία. ηλεκτρονικές ε, πληροφορίες για την μεταφορά εμπορευμάτων. Εισηγητής είναι ο κύριο Ντέλη. Κύριε Ντέλη, βλέπω σήμερα είστε όλο χαμόγελα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Συγχαρητήρια κύριε Ντέλη, 47 η ψήφη υπέρ. Και συνεχίζουμε. με τη δεύτερη έκθεση. Ε, προϋποθέσεις όσον αφορά τον έλεγχο για συγκεκριμένες διατάξεις όσον αφορά την απόσπαση των ε, οδηγών στις οδηγές μεταφορές. Κονιέτσουνα είναι η κυρία Συγγήτρια. Η ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Πέρα της οφορίας. Εγκρίνεται. Έχετε πρόβλημα κύριε Μαρινέσκου. <laughs> Allez, nous continuons. Συνεχίζουμε. η την έκθεση για την κινητικότητα, ε, οι ελάχιστε προδιαγραφέ σε σχέση με την ε, μεγίστη διάρκεια οδήγηση σε μερίσια, εβδομαδιαία βάση και ε, χρόνια ξεκούραση και κανόνες για ταχυγραφου Βυρκούνεν είναι η συγκέντρια. ψηφίζουμε. Je ferme le ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε. Έκθεση που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού 1071 του 9 και του 1072 του 9 για να προσαρμοστούν στις εξελίξεις. Συγητής ο κύριος Αρτούγκ. Ψηφίζουμε. Et je ferme le vote. Πέρασε. Εγκρίνεται. Et nous continuons les votes, s'il vous plaît. Συνεχίζουμε τις ψηφοφορίες, τρόπο ψηφίση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας για τις αεροπορικές υπηρεσίες Μαρόκου Ευρωπαϊκής Κοινότητας για να καλυφθεί η προσχώρηση Βουλγαρίας και Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφίζουμε. Le vote est clos. Πέρασε. C'est approuvé. συμφωνία οδικών μεταφορών Γερμανίας και Ελβετίας για την έγκριση ε, κάποιων μεταφορών καμποτάζ με λεωφορεία στις ε, συνοριακές μεθοριακές περιοχές. Ψηφίζουμε. Le vote est Πέρασε ο Με ευρία πλειοψηφία εγκρίνεται. Πρόταση έγκριση προς την Ιταλία για διαπραγμάτευση συμφωνίας με την Ελβετία όσον αφορά κάποιες μεταφορές και καμποτάζ όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταφοράς, τι ε, οδικές και μεταφορά ε, με πούλμαν στις ε, μεθοριακές περιοχές. Ψηφίζουμε. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε στον τη σύναψη συμφωνίας για την αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας της Βόρειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Δομική κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομική Ενέργεια πιο σωστά. Ψηφίζουμε. Le vote. Πέρα τη ψηφοφορία. Σαράντα υπέρ. Εγκρίνεται. Πολύ ωραία. Παρακαλώ. Απαλλαγή. Έκθεση Μοντέιρο. Πρώτα-πρώτα τροπολογίες. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Υπαριθμόν 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πρώτη συμβαστική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, δεν σας το αποτέλεσμα, θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 6 ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να γίνει επαλήθευση για το 15. Ψηφίζουμε για το 15. Πέρα ψηφορίας. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 18. Υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. Ψηφίζουμε για το 18. Πέρας. Το 18 εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Α, αποχές. απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίνεται. Παρακάτω. Έκθεση Γκραπίνη για τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και οργανισμούς. Ξεκινούμε με την υπηρεσία για τη θάλασσα. Πρώτη τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές. Α, απορρίπτεται. Δύο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρία, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τέσσερα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πέντε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται και πάμε παρακάτω αεροπορικές μεταφορές υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται η πρώτη, η δεύτερη υπέρ, κατά α, αποχές εγκρίνεται τρία υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τέσσερα υπέρ, κατά α, αποχές εγκρίνεται πέντε υπέρ, κατά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 ψηφοφορίας. Απορρίπτωτα. 16 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, επαλήθευση για το 17. Ψηφίζουμε. Πέρασε εγκρίνεται. Για τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το σύνολο του κειμένου. Ψηφίζουμε. Πέρασε ο βορείος. Εγκρίνεται άνετα. Και συνεχίζουμε. Με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τους Σιδηροδρόμους. Κοινή Υπηρεσία για τους Σιδηροδρόμους. Πρώτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 8. Ναι, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Θα το επαληθεύσω λεπτονικά. Ψηφίζουμε την τροπολογία 8. Πέρα της ψηφοφορίας. Ναι, υιοθετείτε. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 10. Υπέρ κατά, αποχές, υιοθετείτε. 11 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 12 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 13 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 14 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 15 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψήφο. Ψηφίζουμε. Τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε με πλατιά πλειοψηφία. Συνεχίζουμε. Για το Σεζάρ. Είστε έτοιμοι. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμό 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8. Υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Ξεκινάει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας υιοθετείται. Συνεχίζουμε με το Shift and Rail. Τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ποιος δεν θέλει να ψηφίσει. Υιοθετείτε. Δύο υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τρία υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Έξι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τελική ψηφοφορία. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείται. Συνεχίζουμε με την αεροναυτική και το περιβάλλον. Clean Sky. Τροπολογία 1. Περ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμός 1. Περ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ουφ. Δεν είναι σαφές. Θα το επαληθεύσουμε. Ψηφίσουμε τώρα την 4. Τροπολογία 4. Πέρας ψηφοφορίας. Wow. Υιοθετείτε όμως. Αυτά συμβαίνουν. Συνεχίζουμε. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ορισμένοι δεν ψηφίζετε. Εντάξει, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τώρα να δούμε. Ψηφίζουμε τώρα την 6. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με μία ψήφο. Συμβαίνει και αυτό. 7. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε άνετα. Μπράβο κυρία Γκραπίνη για όλες τις εκθέσεις σας που υιοθετήθηκαν όλες για τις, τους διάφορους οργανισμούς και υπηρεσίες. Συνεχίζουμε. On va vous laisser deux minutes pour ça. Δύο λεφτά σας δίνω για να βγείτε. Ήσυχα όσοι θέλετε να βγείτε. Il, n'est Σταματάμε για 7 λεπτά, συνάδελφοι, γιατί η προσκεκλημένη μας ή ο προσκεκλημένος μας δεν έχει φτάσει ακόμα, άρα έχετε χρόνο για καφέ. 7 λεφτά σας δίνω. Mes ξαναρχίζουμε τις εργασίες μας. Θα συζητήσουμε σε λίγο στη συνεδρίαση με τους συντονιστές την ε, τροποποιημένη δημοσιονομική διαδικασία. Ακριβώς γι' αυτό η γνωμοδότηση που θα συντάξουμε για τους προσανατολισμούς του προϋπολογισμού του 2021 θα είναι η πρώτη συνεισφορά μας στις πρώτες φάσεις της ε, διαδικασίας προϋπολογισμού. Έχουμε σφιχτό χρονοδιάγραμμα, χρονοδιάγραμμα συγγνώμη, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε με το Γενικό Εισηγητή για τον Προϋπολογισμό, τον κύριο Λαγού Τιουγό. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας για να συζητήσουμε το θέμα αυτό του προϋπολογισμού σήμερα. Είσαστε ευπρόσδεκτος και όποτε μας το ζητήσετε η Επιτροπή μας είναι στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε ενδεχομένω τεχνικά θέματα. Είτε εσείς είτε η υπηρεσία σας πρέπει να μας το πείτε αν θέλετε να έρθετε σε επαφή για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Θα σας δώσω 10 με 15 λεπτά για να μας παρουσιάσετε αυτό το γενικό πλαίσιο με μία μικρή εστίαση στα δικά μας θέματα, δηλαδή τις υποδομές μεταφορών και να δούμε πού προχωρήσαμε στον προϋπολογισμό, στις, στους προσανατολισμούς του προϋπολογισμού. Σας ευχαριστώ Α, και καλή χρονιά, έτσι. Ευχαριστώ Καρίμα, ε, καλή χρονιά σε όλους. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Είμαι νέος Ευρωβουλευτής εδώ και έξι μήνες. Ήμουν ασκιώδης εισηγητής στον προϋπολογισμό του 2020 και είμαι γενικός εισηγητής για τον επόμενο προϋπολογισμό του 2021 αν κερδίσουμε 9 δισεκατομμύρια παραπάνω ε, για τον προϋπολογισμό 2020, ε, είναι γιατί κατάφεραν οι πέντε πολιτικές ομάδες ε, συνεργάστηκαν. Είδαν ότι υπάρχει φιλοδοξία από το Κοινοβούλιο με σαφείς στόχους. Συμφωνήσαμε από τον Οκτώβριο και είπα ότι αφού μπορέσαμε να σκεφτούμε, να συνεργαστούμε στο παρελθόν και αν το κάνουμε αυτό και από το Φεβρουάριο και μετά θα είναι πολύ καλό γιατί θα είναι δύσκολη διαπραγμάτευση. Βλέπω ας πούμε ε, ότι στην φιλανδική πρόταση υπήρχε 35% ε, μείωση σε σχέση με αυτό που ζητούσε το Κοινοβούλιο. Αν είμαστε ενωμένοι με σαφείς προτεραιότητες για να εξασφαλίσουμε νέους πόρους δεν θα τα καταφέρουμε εάν δεν ε, συνεργαστούμε. Θα σας δώσω και κάποια στατιστικά και κάποιες γραφικές παραστάσεις Μπορούμε να δούμε τις διαφάνειες παρακαλώ, το PowerPoint. Λοιπόν, να σας πω ποιες είναι οι προτεραιότητες μας. Αφορά και τις μεταφορές. Η πρώτη προτεραιότητα. Θα μιλήσω γαλλικά. Ε, αν μιλάω πολύ γρήγορα, μου το πείτε. Μου το είπα και οι Γάλλοι ότι μιλάω πολύ γρήγορα. Η πρώτη προτεραιότητα είναι να εξασφαλίσουμε το Green Deal. Τη πρόληση μου στη Μαδρίτη. Και όταν βλέπετε τους Μπαγκλαντισιανούς ή τους Αφρικανούς να σας μιλάνε για τα κλιματικά προβλήματα, καταλαβαίνετε, είναι σοκαριστικό. Ε, πέρασα δύο μέρες στον Παμάκο. Ε, εκεί λένε ότι η κλιματική αλλαγή θα προκαλέσει πάρα πολλούς νεκρούς. Και παρά τις διασκέψεις, αν δεν είμαστε ενωμένοι, αν δεν έχουμε σαφείς προτεραιότητες και αν δεν έχουμε μαζί μας τους πολίτες θα τα καταφέρουμε. Ε, ο παλιός ε, Γάλλος πρωθυπουργός της δεξιάς ε, που ήταν πρόεδρος της Αρμόδιας Επιτροπής είπε ότι οι υπουργοί συζητούσαν, α πούμε, αλλά κάθε φορά πίεζαν για να μην υπάρχει καμία υπέρβαση. Θα πρέπει λοιπόν το Κοινοβούλιο να είναι σαφέ, σαφές, με σαφεί στόχου, ε, και τους πολίτες μαζί για να εξασφαλίσουμε περισσότερους πόρους από τους υπουργού. γιατί αλλιώς θα μας κόψουν τα φτερά. Ε, λοιπόν, το, τα κλιματικά είναι πολύ σοβαρά και παρά τις διεθνείς διασκέψεις ε, η αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι τρι, προ, τρεις φορές μεγαλύτερη από τις δεκαετία του 60. Το πρόβλημα επιδεινώνεται Έχουμε φτάσει στο σημείο το μη παρέκει. Ε, οι κλιματολόγοι σας βλέπουν αυτή την, ε, τη γραφική παράσταση. Ε, βλέπετε το μπλε, ας πούμε, με, που δείχνει πώς εξέλιξονται ε, οι παγετοί. Ε, το 20% ε, είχαμε παλιότερα, κατά μέσο όρο, που έλειωνε τον Ιούνιο. Τώρα λιώνει το 40 45% τον Ιούνιο. Α, φτάνουμε στο μη παρέκει. Στη Μαδρίτη Απογοητευτήκαμε. Όλα τα κεφάλια στρέφονται με ελπίδα προς την Ευρώπη. Είχαμε μία ε, ομάδα, ε, δύο εβδομάδε που κάνει ωραίε συζητήσει, φιλόδοξες κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά για τις μεταφορές. Εάν θέλουμε τα δέκα επόμενα χρόνια να μειώσουμε δια δύο το διοξίδιο του άνθρακα, θα πρέπει να αμονώσουμε τα, τα κτίρια, τη γεωργία κτλ. Ε, τα πιο δύσκολα και δαπανηρά προβλήματα είναι πώς θα αμονώσουμε τα κτίρια, πώς θα ασχοληθούμε με τις μεταφορές και το θέμα της γεωργίας. Γι' αυτό λοιπόν ε, στρέφομαι προς εσάς, ε, πρέπει να, βρείτε, να βρούμε συμμάχους ε, στο Κοινοβούλιο. 40 χρόνια, δεν πρέπει μπορούμε να περιμένουμε, τώρα πρέπει να δράσουμε. Ε, πριν από τα Χριστούγεννα, μα, είδαμε τους αρμόδιους, μας είπαν στις 14 Ιανουαρίου ε, θα βγει ένα νέο έγγραφο, αλλά δεν υπάρχει νέο χρήμα. Ε, υπάρχει απογοήτευση. Ήταν δύο, αυτούς τους δύο συμβούλους ε, μας είπαν ότι δεν υπάρχει ε, πολλά, πολύ φρέσκο χρήμα, 7 δισεκατομμύρια για 7 χρόνια, δεν είναι πολλά. Ε, θέλουμε λοιπόν να προωθήσουμε τις δράσεις με τους πολίτες, αλλά πρέπει να ασκήσουμε πίεση. Χρειαζόμαστε πίεση του Κοινοβουλίου και των πολιτών. Αν διαβάσατε αυτό το έγγραφο της περασμένης εβδομάδα, η, η νέα Κομισιόν λέει ότι λείπουν χρήματα. Η παλιά Κομισιόν είχε ένα λιγότερο φιλόδοξο ε, πρόγραμμα, έλεγε ε, τα λείπανε ας πούμε 215 ε, δισεκατομμύρια ε, ευρώ κάθε χρόνο. Ε, μην, και μην ξεχνάμε και το κοινωνικό κόστος και τις πολιτικές προσαρμογής. Αυτά τα λέγει η παλιά Επιτροπή. Και αν θέλουμε να επιταχύνουμε και να μειώσουμε δια δύο το διοξείδιο του άνθρακα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα κοινωνικά στοιχεία ε, και λείπουν σε αυτήν την περίπτωση 500 εκατομμύρια. Έτσι. 500, συγγνώμη, δισεκατομμύρια. Το πιο σημαντικό θέμα είναι αυτό. Απέναντι σε αυτές, ε, σε αυτές τις ανάγκες 270 με 300 δισεκατομμύρια ας πούμε, που λείπουν. Ε, τώρα τι μας δίνουν 6 δισεκατομμύρια ας πούμε. Ελπίζουμε να φτάσουμε στα 16. Η τράπεζα του κλίματο ε, δεν θα δώσει τίποτα περισσότερο όμω. Ε, σε ό,τι αφορά το φρέσκο χρήμα, είναι αυτά τα 7 ε, δισεκατομμύρια για 7 χρόνια. Δεν είναι τίποτα, θα πρέπει να προχωρήσουμε. Η Καρίμα είπε ότι πρέπει να τα ξαναπούμε εκτό από σήμερα. Θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα project, τι ανάγκε των χωρών, τι ανάγκε για ε, υποδομέ, την καθημερινότητα, στι μεταφορέ να έχουμε του πολίτε στο μέρο μα για τι χρηματοδοτικέ ανάγκε. Και στον τομέα του, των οικοδομών τα πράγματα είναι α, σαφή. Τα δέκα επόμενα χρόνια θα πρέπει να μονώσουμε τα μισά κτίρια. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, δεν είναι περίπλοκο. Αν έχουμε τα μέσα θα το κάνουμε. Στον τομέα των μεταφορών πρέπει να σκεφτούμε και να κοινοτομήσουμε. Ξέρετε ότι διαπραγματευόμαστε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Διαπραγματευόμαστε τον προϋπολογισμό του 2021, το, την Πράσινη Συμφωνία και το Πουδουπού. Και για τον προϋπολογισμό του 2021 ε, πρέπει να τον δούμε στο πλαίσιο του Πουδουπού. Μια νέα κρίση μίλησα με τον Νίκολα Σμιτ για τις κοινωνικές υποθέσεις επίτροπο, είναι ότι κατά διάρκεια της, ε, ε δική μα θητεία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την κλιματική κρίση, να συνεχίσουμε τι κλασικέ πολιτικέ και να αντιμετωπίσουμε και νέα οικονομική κρίση. Η χρηματοπιστωτική κρίση. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τη βασική αποστολή τη Ευρώπη, να αντιμετωπίσουμε μια ιστορική πρόκληση. Για πρώτη φορά στην ιστορία τη ανθρωπότητα θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κλιματική κρίση και οι περισσότεροι οικονομολόγοι θεωρούν ότι θα έχουμε και μια νέα οικονομική κρίση. Ε, αυτό είναι το συνολικό χρέο των ΗΠΑ. Ε, ιδιωτικό δημόσιο. 2.500 ε, ε, δισεκατομμύρια. Αυτό είναι της Κίνας. Ε, μιλάμε τώρα για ένα αεροπλάνο ουσιαστικά ε, με τους δύο κινητήρες προβληματικούς, ΙΠΑ και Κίνα. Έτσι. Δεν είδαμε ποτέ τέτοια εξέλιξη του χρέους ε, σε αυτές τις δύο χώρες. τελευταία φορά το 2007 που είχαμε ε, κερδοσκο... κρίση, είχαμε κερδοσκοπία 14 δις. Τώρα έχουμε φτάσει στα 39. Δηλαδή το επίπεδο της κερδοσκοπίας σήμερα στις χρηματαγορές είναι δυο φορές πιο ψηλό, δυο φορές χειρότερο από το 2007. Τώρα είναι κάθε μήνα το, το που προσοχή έχουμε μια νέα, εγκυμονείται μια νέα ε, κρίση, ε, πολύ πιο ε, έντονη από αυτή που είχαμε το 2007. Ε, γι' αυτό μιλάμε για ένα σύστημα α, αντασφάλισης της απασχόλησης. Ε, αντί να απολύουμε τους ανθρώπους ε, αν υπάρχει πρόβλημα, ε, να μειώσουμε το χρόνο εργασίας, να κρατήσουμε το, το χρόνο, να κρατήσουμε συγγνώμη τον κόσμο όμως. Είδα λοιπόν την Νίκολα Σμιτ και το συζητήσαμε. Δεν σας αφορά τόσο πολύ, αλλά οι δύο βασικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου είναι να χρηματοδοτήσουμε την Πράσινη Συμφωνία με ένα τεράστιο κομμάτι για τι ε, μεταφορέ και να προστατεύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του εργαζόμενου από την επόμενη χρηματοπιστωτική κρίση. Δεν ξέρω αν θα ξεσπάσει τώρα ή του χρόνου. Ε, ρωτήσαμε 200, 230 οικονομολόγους και οι περισσότεροι είπαν ότι θα ξεσπάσει το 2020. Αλλά όπως είπε και ο Κέννεντι, καλύτερα να μας το ρέψουμε και να διορθώσουμε τη στέγη όταν ο καιρός είναι καλός παρά να περιμένουμε τη βροχή. Θα πρέπει λοιπόν να χρηματοδοτήσουμε την Πράσινη Συμφωνία σε όλη την επικράτεια και να προετοιμα προετοιμαστούμε για την επόμενη κρίση και να μειώσουμε τις επιπτώσεις για τους εργαζόμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν πόροι. Ε, μιλήσαμε με τον πρόεδρο της τράπεζας Bay ε, και την τράπεζα του κλίματος, η οποία όμω μπορεί να μας δώσει μόνο 16 δις επιπλέον. Και ποτέ η, ε, ε δεν είχε προβλέψει τόσο χρήμα Αυτό σα αφορά γιατί στι μεταφορέ υπάρχουν μακροπρόθεσμες, γίνονται μακροπρόθεσμες επενδύξεις ε, που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από μια τράπεζα κλίματο αν έχει τα μέσα. Αν δεν υπάρχουν επιπλέον πόροι, ε, τι θα σα πω, ότι η ΕΚΤ ας πούμε δεν έχει δικαίωμα να, έχει, να είναι μέτοχο στην τράπεζα κλίματο και η ίδια η τράπεζα κλίματο έχει γελία, γελίους πόρους. Αν είχε πραγματικά πόρου, θα άλλαζαν τελείω τα πράγματα. Ε, γιατί θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει αυτή η τράπεζα και τις ε, υποδομές μεταφορών. Ε, η ΜΠΕΙ, λοιπόν θα έχει μια θηγατρική, την τράπεζα κλίματος. Στην Επιτροπή Προϋπολογισμού τις επόμενες, αρχίζουμε τις ακροάσεις την επόμενη εβδομάδα για όλα αυτά τα θέματα που σα ανέφερα, γεωργία, ε, μόνο των κτηρίων κτλ. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε νέου πόρου. τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν μπορούν να βάλουν στον κουμπαρά 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Θα πρέπει... Εδώ βλέπει πώς, πώς εξελίσσονται τα μερίσματα στην Ευρώπη. Υπάρχουν ε, κέρδη, οι εταιρείε θα πάνε καλά. Θα πρέπει να δούμε πού πάνε αυτά τα κέρδη. Ε, τα μοιράζονται με τους ε, εργαζόμενους, κάνουν επενδύσεις ή απλώς γίνονται μερίσματα στις τσέπες των ε, μεγάλων, ας πούμε. Ε, στην πραγματικότητα, όταν οι τράπεζες αυτές δεν την πραγματική οικονομία, αυτό είναι πρόβλημα. Ε, όταν ήταν πρόεδρος ο Ντελόρ, τον είχα συναντήσει και έλεγε ότι αν συνέχιζε την, ε, την, ε, το φορολογικό ανταγωνισμό, οδεύει προς την καταστροφή. Εδώ έχουμε πάρα πολλά κέρδη, αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε για την έρευνα, για τις υποδομές. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα. Ε, ορισμένοι λένε ότι αν είχα περισσότερα, ας πούμε 5 δισεκατομμύρια περισσότερο για τις ε, για την έρευνα θα ήταν αλλιώ τα πράγματα. Βλέπετε τι γίνεται στην ε, Ευρώπη εδώ και τι γίνεται στην Αμερική. Ε, από το Ρούσβελτ μέχρι το Τραμπ ο, ο φόρος είναι 38%. Ενώ στην Ευρώπη είμαστε στο 19%. Ε, μας μιλάνε για το New Green Deal. αυτό παραπέμπει στις ΗΠΑ και στο New Deal. Ε, ο οποίο Ρούσβελτ μάλιστα δημιούργησε ένα νέο φόρο τότε για να έχει περισσότερα έσοδα. Εδώ έχουμε, αναφέρθηκαν ε, κάποιοι στον Κέννεντι ας πούμε. Ε, ο Κέννεντι όμως έκανε πολλά πράγματα. έδωσε περισσότερα λεφτά στην NASA ας πούμε, τα πολλαπλασίασε επί 15. Ενώ ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός αυξήθηκε επί 3. Ο έλεγε ότι μπορούμε να πάμε στο, στο φεγγάρι, δεν χρειαζόμαστε τους σπόρους. Αυτά. Ποια είναι η άποψή σας για το 2030, για το 2050, ε, με βάση την ε, φιλοδοξία του New Green Deal που θέλει να μειώσει δια δύο, να διαιρέσει δια δύο τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, τι project έχουμε στο τραπέζι και δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε. Πρέπει να πιέσουμε τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Βλέπουμε στην Γερμανία και στη Γαλλία ε, και στην Ιταλία προγράμματα τα οποία δεν προχωράνε όμως και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Μήπως πρέπει να έχουμε νέους, ε, νέα εργαλεία, ε, νέο προπολογισμό. Θα πρέπει να έχει περισσότερα λεφτά η Τράπεζα Κλίματος. Τι έχει ο προπολογισμό και τι υπάρχει εκτός προπολογισμού. Μπορούν να μας βοηθήσουν γιατί εγώ δεν ξέρω και πολλά. α τα πούμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Ας δούμε τις πραγματικές μας ε, ανάγκες, ας δούμε τις επιπτώσεις ε, στην απασχόληση, ας δούμε τι εργαλεία χρειαζόμαστε. Ζητώ συγγνώμη που είπα τόσα πολλά. Ε, ήμουνα σύμβουλος επί πολλά χρόνια. Τις επόμενες ε, τρει εβδομάδε έχουμε τις διαπραγματεύσει. Πρέπει να σκεφτούμε τη θέση μα. Πολύ πλήρης η ομιλία σας κύριε Λαροτόρο και τώρα να συζητήσουμε. Πρώτος ο κύριος Μαρινέσκου για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση αυτή για την παγκόσμια οικονομική κατάσταση. Εδώ είναι η Επιτροπή Μεταφορών όμως. Και θέλουμε να μας πείτε Πώ προτείνεται να οικοδομήσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προπολογισμό του επομένου έτους ε, χωρίς ε, πι δελτα πι. Γιατί για την ώρα δεν προβλέπεται κάτι και ταυτόχρονα χωρίς ε, κάποια πρόταση από την Επιτροπή Περιπολογισμού. Για να εξηγήσουμε λοιπόν λίγο τη νέα διαδικασία, γιατί είναι νέα διαδικασία και οι συνάδελφοι θα θέλουν φαντάζομαι να την μάθουν. Λοιπόν, ξανά. Άκουσα εδώ πέρα για Κέννεντι, διάφορα πράγματα για τη Γαλλία, αλλά τι ε, περιμένετε ε, από την επόμενη πρόταση του προπολογισμού, του Κοινοβουλίου για τον προπολογισμό για τον προπολογισμό του 2021. Τι θέλετε από τις οριζόντιες επιτροπές. Πώς θέλετε να είναι η έκθεσή σας, τι θέλετε να γράψετε. Υπάρχουν δύο πράγματα. Νέες πολιτικές που θα ξεκινήσουν. Εάν εγκριθεί το ΠΔΠ, ίσως όχι, οπότε τότε θα έχουμε έναν μεταβατικό προπολογισμό και οι πολιτικές θα οι υφιστάμενες που μπορούν να συνεχίσουν, αλλά τρία χρόνια όπως ξέρετε. Υπάρχουν πολιτικές που θα συνεχίσουν για άλλα τρία χρόνια. Πώς έχει η κατάσταση με το Brexit. Το Ενωμένο Βασίλειο ε, θα πρέπει να πληρώνει, αλλά τρία χρόνια είναι ή όχι. Ε, αυτά πρέπει να μας απασχολούν. Αυτά απασχολούν εμένα τουλάχιστον και θέλω να μάθω την άποψή σας. Τώρα εντάξει τα υπόλοιπα. Καλά, αλλά πείτε μας ποια είναι η αποψή σας για τον προϋπολογισμό της κοινότητας ε, του επομένου έτους. Ευχαριστούμε κύριε Μαρονέσκου. Κυρία Γκαρθία Μουνιός, ευχαριστώ κύριε Λαρουτούρου για την ε, παρουσίασή σας. Εμείς στην Επιτροπή Μεταφόρων ενδιαφέρομαστε πάρα πολύ για αυτές τις ε, συνομιλίες για τον ε, προπολογισμό. Είναι πάρα πολύ βασικό θέμα για την συνδεσιμότητα, την συνοχή, ε, τα κοινωνικονομικά της Ένωσης και τη συνοχή τους. Αυτά τα μέτρα πρέπει να είναι συγκεκριμένα για να προσφέρουν αυτό στους πολίτες. Ακριβώς όπως η ελεύθερη διακίνηση αγαθών και πολιτών και προσώπων. Χρειάζεται ε, μεταφορές, χρειάζεται υποδομές η Ευρώπη και εδώ κλειδί είναι οι μεταφορές. Άρα θα πρέπει να κάνουμε βήματα πρόοδου για περισσότερη βιωσιμότητα για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους για την κλιματική αλλαγή και για το πράσινο σύμφωνο. Ε, αυτό που είπατε ε, ακριβώς το μέσο χρηματοδότηση είναι πολύ σημαντικό και προτεραιότητα για την ε, μετάβαση. Οπότε έτσι θα πρέπει να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτή την ευφυή την βιωσιμή και με ασφάλεια την οποία και θέλουμε. Και επίσης εκεί πρέπει να γίνουν οι επενδύσεις καινοτομία, βοήθεια στην τεχνολογία όπως η τηλεματική ε, αναζήτηση εναλλακτικών καυσίμων, ε, συνδυασμένες μεταφορές, με, μετακίνηση μεταφοράς εμπορευμάτων προς το σιδηρόδρομο, όλα αυτά μας ενδιαφέρουν στη δική μας πολιτική ομάδα τους σοσιαλδημοκράτες. Όλα αυτά θέλουμε να γίνουν προτεραιότητες του προϋπολογισμού και τονίζουμε αυτή την ευκαιρία το ότι πρέπει η πρόταση της Επιτροπή μας να προωθηθεί όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Κύριε Ρικέ, είτε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιέρ, ευχαριστούμε για όσα μας είπες. Θέλω να σταθώ σε κάποια σημεία που δεν αφορούν τα δημοσιονομικά με τη στενή έννοια. Πρώτον, γνωρίζουμε ότι χρειάζονται επενδύσεις και πολύ και για την κλιματική αλλαγή και για την οικονομία της εσωτερικής αγοράς και για την ε, ε, οικολογική μετάβαση πρέπει να είναι και η οικονομική. Να μην έχουμε προϋπολογισμό λιτότητας. Μην πάνε αλλού οι επενδύσεις. Άρα Αλλαγέ πρέπει να γίνουν και στα χρηματοοικονομικά και πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε τα απαραίτητα, όχι τα ευκταία, τα αναγκαία νούμερα. Και στέκομαι στο εξή ακόμα και αν υπήρχαν τα αναγκαία κεφάλαια για τις αναγκαίες επενδύσεις, οικονομικά, κοινωνικά, για, το, την κλιματική αλλαγή, χρειάζεται να μην έχουμε τόση γραφειοκρατία για τις επενδύσεις για να μπορεί να υπάρχει εύκολη αδειοδότηση. Γιατί τώρα η, μέση όρη, ο μέσος όρος τέλο πάντων από έγκριση σε υλοποίηση είναι 7 χρόνια. Και μιλούμε για επενδύσεις από πλευράς πρακτικής. Μην καταντούμε να υλοποιείται αυτή η επένδυση με το επόμενο δημιουργικό πλαίσιο και συμφωνώ ότι θα πρέπει σύντομα να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία όλων αυτών. Να μην έχουμε τόσους φραγμούς και πρόσβαση στην πίστοση. Γιατί ακόμα και αν είχαμε τα μέσα τα οικονομικά δεν έχουμε τα διοικητικά ούτως ώστε να πάμε στις επενδύσεις. Είναι θέμα επικουρικότητας. Οπότε ακόμα υπάρχουν πολλά προβλήματα. Επομένως θα πρέπει και στο μέτωπο της γραφειοκρατίας να δοθεί μάχη, όχι μόνο στον προϋπολογισμό. Ακόμα και αν υπάρχουν τα αναγκαία χρήματα δεν μπορούμε εμπρόθεσμα να τα καταφέρουμε. Κοφ. Ε, ευχαριστώ. Ε, εμένα μου άρεσε η παρουσίαση. Ε, καλό είναι πάντα να εξετάζουμε το ιστορικό πλαίσιο, να συνειδητοποιήσουμε ότι 90 χρόνια πριν είχαμε το New πριν από 60 χρόνια ξεκίνησε η αποστολή προς τη Σελήνη, πριν από 30 χρόνια έπεσε το τείχος του Βερολίνου. Οπότε βλέπουμε ανά τρία κοντά αιτία ε, τις εθνικές κυβερνήσεις και την ε, διεθνή συνεργασία για να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις. Το ίδιο πνεύμα χρειαζόμαστε και τώρα. Η πρόκληση νομίζω είναι και ήταν αυτό σε κάποια από τα γραφικά σας τα υπερκέρδη κάποιων εταιριών. Πώς θα τα πάρουμε αυτά τα λεφτά. Υπάρχουν αυτά τα λεφτά και οπωσδήποτε αν δει κάνει ε, την Ευρωπαϊκή Τραπεζα Επενδύσεων και άλλα θεσμικά όργανα είναι διατεθειμένοι να χρηματοδοτήσουν το πράσινο New Deal. Απλά θέλουν την ουσία του τι είναι αυτό το New Deal. Θα μπορούσε παραδείγματος χάρη να είναι ένα πρόγραμμα ανακαίνησης των μισών σπιτιών μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επένδυση στις εφόρες ε, μεταφορές. Εμείς λοιπόν πρέπει να βρούμε αυτά τα έργα και καθώς διευρύνεται η Ένωση ε, στα νοτιοανατολικά να γοητεύσουμε και αυτούς που θα λάβουν τις αποφάσεις ε, να πούμε ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από τα ορυκτά κάψιμα, να πάμε στις ανανεώσιμες, να υπάρξουν βελτιώσεις στον σιδηρόδρομο, στις θαλάσσιες μεταφορές που είπαμε πριν, αλλά πρώτα απ' όλα υπάρχει μια συζήτηση του να πείσουμε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις και να υπάρξει αυτή η χρηματοδότηση. Πρέπει όμως να είμαστε φιλόδοξοι και νομίζω πως αυτά τα οποία είπατε μας δείχνουν πόσο μεγάλη πρόκληση αντιμετωπίζουμε. Και η ομορφιά του Ευρωπαϊκού Πράσινου Deal ε, και των σχετικών επενδύσεων είναι ότι είναι μια σταθερή μορφή επένδυσης για τα επόμενα 30 χρόνια. Δεν είναι κάτι στο γόνατο ε, που θα εξαφανιστεί. Πρέπει να υπάρξει μια συνεχής όθηση για να γίνει αυτό το πράγμα. Για τις επενδυτικές τράπεζες ε, και τις εθνικές ε, κυβερνήσεις είναι πιο εύκολο έτσι να προγραμματίσουν από ότι για κάποιες άλλες προκλήσεις πριν από 30, 60 και 90 χρόνια. Σας ευχαριστώ. η κυρία Σαμπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί εδώ και χρόνια τρόπου μεταφορών και υποδομών που είναι υπεύθυνε ε, για την απορρίθμιση του, κλι, κλίματος. Ο φόρος, α πούμε, για την κυροζήνη στα αεροδρόμια ε, και η χρηματοδότηση νέων αυτοκινητοδρόμων. Ε, πριν από λίγο καιρό ε, είπαμε ότι υπάρχει κλιματική και περιβαλλοντική επίγουσα ανάγκη. Ε, ο προπολογισμό είναι ένα εργαλείο για να διορθώσουμε την κατεύθυνσή μα και να μειώσουμε το διοξείδιο του άνθρακα στι μεταφορέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θέσει τέλο στη χρηματοδότηση μεγάλων περιττών project μέσω ενό μηχανισμού αλληλοσύνδεση των μεταφορών στην Ευρώπη. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Τον αυτοκινητόδρομο ε, μεγάλη ε, παράκαμψη ε, στα δυτικά τη Ευρώπη. Πού μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πρωταθλητέ στην καταπολέμηση ε, Τη αλλαγή του κλίματο όταν δίνουμε α πούμε σε μια εταιρεία 163 εκατομμύρια για να φτιάξει αυτό το μεγάλο, τη μεγάλη παρακαμπτήριο στα δυτικά που είναι αυτοκινητόδρομο παρακαμπτήριο. Θα πρέπει να πάμε προ τι μικρέ συνδρομικές γραμμέ, γιατί ενώ αυτή τη στιγμή που έχουμε αυτό το πρόβλημα, στην πραγματικότητα κλείνουν πολλοί σιδηρόδρομοι, πολλέ γραμμέ σιδηροδρομικέ και ειδικά τα τρένα νύχτα. Ε, αυτά μα εξασφαλίζουν όμω τη σύνδεση των διαφόρων περιοχών. Θα πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση σε δημόσιε μεταφορέ ε, ίσως να μας πείτε ότι δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει να, αυτές οι μεταφορές να είναι δωρεάν. Ένα μέτρο θα ήταν ε, κοινωνικά δίκαιο και κλιματικά δίκαιο. Αυτά ευχαριστώ. Τον εισηγητή και την πρόεδρο. Κυρία Μοντερό, έχει το λόγο. Muito obrigada, Presidente. Agradeço ao, ao, colega, ao colega... Ευχαριστώ, Πρόεδρε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λαρουτούρου. Μας έδωσε μια πρώτη δόση διευκρινήσεων. Επίσης, συμφωνώ και με τον κύριο Μαρινέσκο σε σχέση με το τι περιμένουμε, τι προσδοκούμε. Θέλουμε χείρα βοηθείας για να μπορέσουμε όλη αυτή την ε, διαδικασία του προϋπολισμού του 2021 να την πλαισιώσουμε και σας υπενθυμίζω ότι αφού μιλάμε για κλιματικές επιπτώσεις, ε, περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ. θα πρέπει να προσέξουμε όλα εκείνα τα σημεία που έχουν θεμελιώδη σημασία για την Ένωση. Όμως όλα αυτά δεν είναι κάτι το νέο. Επίσης πρέπει να σας πω ότι εδώ είναι Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Ο δε τουρισμός καλύπτει και ένα σωρό κλάδους που θα πρέπει να μην τους ξεχνούμε. Ταξίδια, τουρισμός, όλα αυτά αυξήθηκαν τελευταία. Πρόκειται για εκρηκτική αύξηση της δραστηριότητας. Ας πούμε όταν κάποιος μιλάει για τη Γεωργία και εκεί ε, θα πρέπει κανείς να σκέφτεται τον τουρισμό δημιουργεί επίσης πάρα πολλές ε, εξαγωγές. Επίσης με τον βιώσιμο τουρισμό έχουμε δημιουργία απασχόλησης και να μην ξεχνάμε ποιος είναι ο στόχος μας. Βιώσιμος τουρισμός, εφής, προορισμοί, νήσι κλπ. Άρα θα πρέπει προς τα εκεί να προσπαθήσουμε και αποτελεσματικά. Οπότε για πέστε μας, εσείς για τον επόμενο προπολογισμό της χρήση του 2021 θα λάβετε υπόψη τον τομέα αυτών. Μπορείτε να προτείνετε συγκεκριμένες δράσεις, γιατί αυτό περιμένουμε. Κονδύλι για τον βιώσιμο τουρισμό. Είναι πιθανό, τι λέτε. Μπορούμε να το καλύψουμε και αυτό στις διαπραγματεύσεις που ακολουθούν. Μπορείτε να μας το υποσχεθείτε, γιατί έτσι θα βοηθήσετε τη δουλειά μας. Είναι σημαντικός ο τομέας για όλες τις περιφέρειες και όλη την Ευρώπη. Κύριε Παρνιά, ευχαριστούμε κύριε Λαρουτούρου για όσα μας είπατε. Είναι οικονομικό το θέμα και μεγάλη πρόκληση το Green Deal να τύχει χρηματοδότησης. Επίσης δεν πρέπει να ξεχάσουμε κανέναν τομέα, να υπάρξουν επενδύσεις και να σταματήσουμε να δίνουμε πενταροδεκάρες. Εμείς οι πράσινοι εδώ και χρόνια στην Επιτροπή αυτή λέμε ότι ο σιδηρόδρομος θα πρέπει να ενισχυθεί. Μπορεί να φτιάξει απασχόληση και να μειώσει τις βλαπτικές εκπομπές επενδύσεις σε βασικά έργα υποδομής στις μεγάλες γραμμές. Και εκεί που δεν έχουμε πολύ κόσμο, αλλά και στα ψηφιακά. Τα συζητήσαμε και σήμερα το πρωί και για τις αλλαίσεις μεταφορές. Προς, προς τα εκεί να προσπαθήσουμε. Αλλά και ο βιώσιμος τουρισμός θα πρέπει να καλυφθεί. Ναι, να φορολογηθεί το κέρδος, αλλά αυτό τώρα είναι παλιά ιδέα, αλλά δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Αν δεν το κάνουν αυτό τα κράτη, θα πρέπει να ενεργήσει από αυτό το κοινοβούλιο. Χρειάζεται νέο ταμείο, πρέπει να επιστρατεύσουμε τις επιχειρήσεις για αυτή την μετάβαση ξεκάθαρα στάνταρ μέσω μακροπρόθεσμα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα του περιβάλλοντος. Να αλλάξουμε την κατασκευή τη βιομηχανική των μηχανών και να έχουμε αυστηρή νομοθεσία για την κερδοσκοπία. Έχουμε το πράσινο σύμφωνο, αλλά πρέπει να προσέξουμε τι γίνεται με οδικές μεταφορές σε σχέση με σιδηροδρομικές. Στο Invest EU καλύπτονται κάποια κριτήρια συνοχής, γιατί δεν υπάρχει συνέπεια με τους κλιματικούς στόχους. Θα πρέπει ειλικρινά να δούμε πώς καθορίζονται, πώς ορίζονται αυτά τα κριτήρια γιατί για το κλίμα θα πρέπει να ευνοήσουμε κάποιες λύσεις και κάποιες όχι. Να σταματήσει η χρηματοδότηση κάποιων ε, κινήσεων που είναι κακές για το κλίμα. Ο ε, Πρόεδρος, σας ευχαριστώ κύριε Παρνιά. Για κοιτάξτε κάτι άλλο που για μένα είναι σημαντικό. Η Επιτροπή των Προϋπολογισμών έχει κάποια θέση, όπως και το Κοινοβούλιο, για αυτό το Ταμείο Μετάφρασης, 4,8 δις και τελικά 5,7 είπε η Κομισιόν. 5,7 δις. Καλό, θα βοηθήσει κάποιες περιφέρειες που θα πρέπει να μπουν στο παιχνίδι της ενεργειακής μετάβασης. Αλλά θα πρέπει αυτό να συνδεθεί με τα εθνικά προγράμματα. Τα ενεργειακά. Τι θα κάνετε, θα προσαρμοστείτε, θα πιέσετε σε επίπεδο προϋπολογισμού για τα εθνικά προγράμματα. Άλλο. Λέει 10 δις κύριε κυρία Φόντερ Ναι, ναι, δεν είναι αυτά για τη μετάβαση κύριε Λαροντρού. Τι, ένα, τρεις, πού να το βρούμε. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε τους ίδιου πόρου. Λέμε για φόρους, πολλά. Για το σύνολο των μεταφορών θα πρέπει η Κομισιόν να δει τι γίνεται με την Ευρωβινιέτα, το σήμα. Εάν προσπαθήσει ένα κράτο μέλος, Τι θα είναι αυτό, εθνική πολιτική ή όχι. Άρα, γι' αυτό σας λέω. Ο προϋπολογισμός επίσης θα πρέπει να βοηθάει στην, στην καινούργια στάθμιση των πραγμάτων στις μεταφορές. Και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να γίνει αυστηρή για την επιλογή των έργων και προγραμμάτων. 25% είναι οι επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση. Όμως, ε, ο στόχος είναι 50% για την κλιματική αλλαγή. Άρα, 25 ή 50. Κάτι πάει στραβά. Τελευταίο δε. Θα πρέπει να προσέξουμε τις προσαρμογές. Κανένας δεν το προσέχει αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιο ταμείο σήμερα. Γιατί η επανάσταση δεν είναι μόνο η ψηφιακή, είναι και η οικολογική. Τι γίνεται με τη βιομηχανία αυτοκινήτων, τι γίνεται σε κάποια σημεία της Γερμανίας, κλείνει ένα εργοστάσιο, πεθαίνει όλη η περιοχή. Μπά και έρθει ο λόγος, η ώρα, συγγνώμη, να κάνουμε αυτό που πρέπει. Και να θεσπίσουμε κάποιο κονδύλιο, ας πούμε, για την προσαρμογή όχι για το Brexit, αλλά για την κλιματική αλλαγή. Γιατί ξαφνικά μπορεί να ανακύψουν καταστάσεις, οπότε θα χρειάζονται κάτι τέτοιο κάποιοι τομείς και όχι κάποιοι άλλοι. Μήπως μπορούμε να αρχίσουμε προσπάθεια πάνω σε αυτό και για τους ίδιους πόρους επίσης να υπάρχει συγκεκριμένος άξονας. Μιλάμε για φόρους και μιλάμε για κάποια πλεονεκτήματα που γίνουν όλοι κερδισμένοι κύριε Λαρουτούρου. Πολλές είναι οι ερωτήσεις. Και σας δίνω το λόγο να απαντήσετε. Απαντάω στο τελευταίο ερώτημα, αν μπορούμε να συνεργαστούμε. Είμαι εδώ σήμερα. Γιατί, γιατί έχω όρεξη να συνεργαστούμε. Έχω πέντε εμπειρογνώμονες ε, στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Θα μπορούσα απλώς ε, κλασικά να κάνω, να επιλέξω ας πούμε τις καλύτερες ιδέες σας, τα best of ας πούμε. Αλλά όχι, ήρθε εδώ. Εγώ που είμαι ευρωβουλευτής προσπαθώ να έρθω σε επαφή με τους γέρους, τους γέροντες, τους σοφούς γέροντες που μου έδωσαν ε, οι συμβουλές. κύριε Μαρινέσκου, έχετε την αίσθηση ότι χάνετε ε, το χρόνο σας, ζητώ συγγνώμη, αλλά ε, ακούσαμε από ένα παλιό υπουργό ότι το Κοινοβούλιο δεν θα κερδίσει τίποτα εάν δεν έχει μαζί του τους πολίτες αυτή τη διελκυστίνδα με το Συμβούλιο. Η Επιτροπή Προπολογισμού δεν, δεν ξέρει αυτά που ξέρετε εσείς για τι μεταφορέ. Ήμουνα, είμαι, σύμβουλο για 11 χρόνια. Θα μπορούσα να το παίξω επαείοντα. Αλλά δεν τα ξέρουμε τόσο καλά ε, τα, των μεταφορών. Είμαστε στην υπηρεσία η Επιτροπή Προπολογισμού, δηλαδή στην υπηρεσία των υπολείπων επιτροπών. Θέλω να δουλέψουμε μαζί. Μπορώ να σα πω τι προτεραιότητε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε ένα προπολογισμό για να φτάσει στο 1,3 του ΑΕΠ. Το λένε όλοι οι συγκητέ. Ε, αλλά αυτό που έλεγε ο Ζαν Αχτουή, που κάθε φορά που ζητάει κάτι παραπάνω το Κοινοβούλιο, οι αρχηγοί πιέζαν, πιέζαν, πιέζαν και ο προπολογισμό εδώ και 20 χρόνια, ο, Πραγματοποιηθεί προϋπολογισμός ε, δεν ξεπέρασε ποτέ το 0,95% του ΕΠ. Έτσι. Θα μπορούσα να κάνω μια σύνοψη όλων των εκθέσεων των εμπειρογνωμών. Αλλά ήρθαμε εδώ πέρα για να κινήσουμε τα πράγματα. Έχουμε μια ιστορική ευθύνη. Η πίεση του κλίματος είναι η πρώτη πρόκληση της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε. Επίσης, οι προτάσεις ε, της ε, Επιτροπής είναι να ε, μειώσουμε κατά 35% το ΣΕΦ, το Connecting Europe Facility και παράλληλα έχουμε φοβερές φιλοδοξίες. Δεν θέλω να τα πω αυτά για να μιλήσω άσχημα για τους Φιλανδούς και τη Φιλανδική Προεδρία. Περιμένετε, περιμένετε λίγο. Το θέμα είναι να υποφεληθούμε από αυτή τη λευκή σελίδα. Η Κομισιόν μας λέει ότι το Φεβρουάριο θα γίνει μια έκτακτη σύνοδος με τους ε, αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Μπορούμε να υποφεληθούμε. Μπορούμε να υποφεληθούμε όλοι από αυτή τη νέα σελίδα που γυρνάει. Δεν μιλάω για τα νομικά εδώ θέματα. Θα διαπραγματευτούμε. Θα μιλήσουμε για το πουδουπού, για το Green Deal και τον προϋπολογισμό του 2021. Ε, μιλάμε και για τους ε, νέους πόρους, νέους ίδιους πόρους. Εμείς ε, θα μπορούσαμε να μπλοκάρουμε το που αν δεν είχαμε προχωρήσει για τους ίδιους πόρους. Θέλουμε με επιχειρήματα να προχωρήσουμε που μιλάνε και πείθουν πολίτες και συνδικαλιστές. Εγώ αυτό που αρνούμε είναι να μας λένε ότι όλα είναι μια χαρά. Θα μειώσουμε το 35% σε σχέση με αυτό που ζητήσατε, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα για το κλίμα και τον πλανήτη, ας πούμε. Εδώ δηλαδή τι είμαστε, μαγικά πράγματα. Μπορούμε να μειώσουμε τις επενδύσει κατά 35% αλλά μας λένε ότι κάνα πρόβλημα για το κλίμα. Συγγνώμη, αλλά ως πολίτης και εκλεγμένος δεν μπορώ να τα εξηγήσω αυτά στους ε, ψηφοφόρους μου ε, τα επόμενα χρόνια. Ε, για το ερώτημα του Ντομινίκ Χικέ, μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν έχω το μαγικό ραβδάκι. Όταν μου λέτε ότι χρειάζονται 7 χρόνια από τη στιγμή που ψηφίσουμε προπολογισμό και την υλοποίηση, το θέμα είναι να μπορούμε να προχωρήσουμε, να κάνουμε προτάσει. Ε, εσείς μας λέτε, να, ε, κυρία Καρύμα, μου λέτε να πιέσουμε εμεί η Επιτροπή Προπολογισμών, το Συμβούλιο. Δεν έχουμε και υπερβολικέ φανταστικέ εξουσίε. Το βασικό είναι να είμαστε αραγέ μέτωπο ε, ως κοινοβούλιο και να κάνουμε κάτι με του ε, ιδίους Δεν πρόκειται να μας δώσει η Ρουμανία, η Γαλλία, η Γερμανία περισσότερου πόρου πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα λεφτά των διαφόρων τραπεζών για το ερώτημα της κυρίας Σαμπή. Ο προπολογισμό δεν μπορεί να διορθώσει την ε, νομική βάση. Δεν είναι η δουλειά του προπολογισμού αυτή. Την άλλη, ε, τις προάλλες ήρθε εδώ ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ε, γιατί είπε ότι θα σταματήσει τις, τη χρηματοδότηση των project με ορυκτά καύσιμα. Θέλουμε κάποιε διευκρινήσει. Και μετά εμείς και η τράπεζα θα μπορούσαμε να δώσουμε μάχη για περισσότερους ίδιους Ε, ο Ντομινίκ Ρικέ είπε ότι ε, η Μπέι δεν μπορεί να είναι μέτοχος στην τράπεζα κλίματος, θα πρέπει να δώσει δικά τη λεφτά. Ε, νομίζω ότι όλα αυτά είναι θεμελιώδη. Αν θέλουμε και προϋπολ... να έχουμε λεφτά και από τον προπολογισμό και εκτό προπολογισμού. Ε, το θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμο για να χρηματοδοτήσουμε μακροπρόθεσμα project. Η 100 δισεκατομμύρια το μήνα έχει η, η ΕΚΤΑ. Η ΕΚΤΑ έχει 2,63. Ε, Όλα τα, τους μήνες υπάρχουν 80 ε, δισεκατομμύρια που φτάνουν στο τραπέζι. Τι κάνουμε με αυτά τα λεφτά. Υπάρχει και η νέα η χρηματοδότηση μέσω Ντράγκη, 20 ε, δισεκατομμύρια, συνολικά 100 εκατομμύρια το μήνα. 1,2 δηλαδή 3 το χρόνο. Τι κάνουμε αυτά τα λεφτά. Το καθεστώς της Κεντρικής Τράπεζας και ο ρόλος της ε, είναι να πολεμήσει για τη σταθερότητα τη σταθερότητα των τιμών. Ε, όταν δεν αφισβητεί τη σταθερότητα των τιμών, θα πρέπει η ΕΚΤ να εξυπηρετήσει και άλλα πράγματα, του στόχου του άρθρου 3 δηλαδή. Στο 3.3 3 μιλάμε για την προστασία του περιβάλλοντο. Θα πρέπει να το υπηρετήσει αυτό το σκοπό η ΕΚΤ. Οι άνθρωποι τη ΕΚΤ λέτε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορεί να αλλάξει γρήγορα την πολιτική τη και να προωθήσει τι μακροπρόθεσμε ε, επενδύσει. Μου λένε ότι έχω άλλα τρία λεφτά. Ε, για την ανάγκη σταθερότητας. Το είπε ο κύριο Κάφ. Ναι, θα πρέπει να δώσουμε κατευθύνσεις και μακροχρόνια χρηματοδότηση. Για το θέμα του Ταμείου μετάβαση, ερώτηση της Προέδρου, είναι εντελώ ανεπαρκέ. Ε, μας λένε ε, και οι Επίτροποι ότι είναι μία απαρχή. Πρέπει να συζητήσουμε με το Κοινοβούλιο, ούτω ώστε να πιέσουμε τους αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων. Το θέμα είναι να έχουμε ε, ιδέες για να προχωρήσει η διαπραγμάτευση. Για τους ίδιους πόρους, για την Ευρωβινιέτα πρέπει να προχωρήσουμε μαζί. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα κάνει μια έκθεση πρωτοβουλία σίγουρα. Θα το συζητήσουμε αύριο στην Επιτροπή Προπολογισμών. Είσαστε ευπρόσδεκτοι, αν θέλετε, να συμμετάσχετε σε αυτέ τι ακροάσει για του ίδιου πόρου, για να έχετε και καλύτερα επιχειρήματα. Γιατί αν μείνουμε με βάση του πόρου που μα δίνουν τα κράτη-μέλη στη διάθεση, που στη διάθεσή μα, δεν θα έχουμε αρκετά λεφτά για το Ταμείο Προσαρμογής. Θα πρέπει να τροφοδοτηθεί και αυτό από ίδιους πόρους. Τι ξέχασα? Pardon. Encore μια νέα σελίδα, ε, διαπραγματευόμαστε έναν ε, ετήσιο προπολογισμό όταν δεν έχουμε καν το πλαίσιο το πολιετέ. Το πού δηλαδή. Είναι μια ευκαιρία για το Κοινοβούλιο, νομίζω. Βλέπουμε ότι οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων είναι μπλοκαρισμένοι. Χθε ήταν ένα σημαντικό ε, πρέσβη, ο οποίο μου είπε ότι αυτή η διαπραγμάτευση είναι σφαγείο. Εμεί μπορούμε να υποφεληθούμε, ούτω ώστε να προτάξουμε τι δικέ μα προτεραιότητε, που είναι σαφεί, για να δούμε τι θα κάνουμε του ίδιου πόρου. Είναι ή να χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά τα project ε, με έναν άλλο τρόπο θα πρέπει να έχουμε ιδέες, να δοκιμάσουμε νέες ιδέες. Θα ξεκινήσουμε τις δικές σας προτάσεις. Είσαστε η πρώτη επιτροπή που επισκέπτομαι είναι πάρα πολύ περίπλοκο αυτό το, τα πράγματα, τα θέματά σας. Ε, θα μπορούσα να έρθω εδώ πέρα με μία στρατιά από επαΐοντες ας πούμε και να κάνω μία σύνοψη των ε, εκθέσεων που βγάλετε τα τελευταία 4-5 χρόνια. Όχι, εγώ θέλω να δουλέψω μαζί πραγματικά. Έχω μέχρι το κράτη ε, επίσημα θα υποβάλω την πρώτη έκθεση ε, σε 15 μέσα, αλλά αυτό δεν είναι ουσιαστικό. Η ουσία είναι ε, θα παιχτεί τον Ιούνιο και Ιούλιο. Έχουμε δηλαδή μερικούς μήνες για να σκεφτούμε μαζί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Είσαστε... Θα σας έχουμε στο πλευρό μας, σύμμαχοι θα μας... σύμμαχους θα μας βρείτε. Έχουμε και εμείς εμπειρογνώμονες, τον κύριο Γικέ, Μαρινέσκου και άλλους που ξέρουν αυτά τα θέματα του προϋπολογισμού. Σας ευχαριστούμε. Ελπίζουμε σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία να μην αφαιθούμε να και ιτηθούμε. Όταν κοιτάμε τον προϋπολογισμό, γιατί ξέρω ότι πήγαμε τον κύριο Ρικέ στο άτυπο υπουργικό, όπου μας είπαν ότι το τμήμα των μεταφορών που έχει προβλεφθεί στον προπολογισμό είναι 9%. Δεν λαμβάνουν υπόψη όμως ότι χωρίς κινητικότητα οι πολίτες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και δείχνουμε εμεί ότι δεν είναι στην πραγματικότητα αυτό το 9% που μας έχουν δώσει. Ε, το ελεγκτικό συνέδριο λέει ότι ο τομέα που πρέπει να δοθούν και να γίνουν οι περισσότερε επενδύσει είναι ακριβώ οι μεταφορέ. Οι μεταφορέ και ο τομέας των ακινήτων, των κτηρίων, ε, των δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ τον ομιλητή μας. Πρώτη συνάντηση αυτή. Το χειροκροτούμε τώρα από αποχωρεί. Notre Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου. 9 η ώρα δύο μέρες, από 9 μέχρι 12.30 και 2.30 μέχρι 6.30 και στις 20 Φεβρουαρίου από τις 9 μέχρι τις 12.30 και τις 3, τις 3 μέχρι τις 6. Προσοχή, προσοχή λοιπόν. Η συνεδρίαση της, στις 28 Ιανουαρίου ακυρώνεται. Σημειώστε στην ε, ατζέντα σας.